Okay. Ευχαριστώ. Euh, Καλησπέρα σα. Λοιπόν, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Ε, θα δούμε καταρχήν την ημερήσια διάταξη και θα κοιτάξουμε να την τροποποιήσουμε. Λοιπόν, οι πολιτικές ομάδες ενημερώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έλαβε άδεια και την άδεια και βέβαια βάσει των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία μια κατεπίγουσα έκθεση για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τις εξωτερικές δράσεις που θα δημιουργηθούν μετά από την επικύρωση σε όλα τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να αποφανθεί για αυτήν ε, την τόσο σημαντική υπηρεσία που θα αποτελεί και τον αντιπρόσωπο η Επιτροπή συγγνώμη, Εξωτερικών Υποθέσεων που θα αποτελεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αποφάσισε και αυτή να συντάξει έκθεση και εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Αύριο θα γίνει η συζήτηση στις συνταγματικές υποθέσεις. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 8 Οκτωβρίου και 19 του μηνός θα περάσει από την Επιτροπή και την επόμενη εβδομάδα θα περάσει από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γνωμοδοτήσουμε για αυτό το θέμα το οποίο αφορά στην θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά ε, ανέθεσαν σε μένα τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τους συντονιστές για την εμπιστοσύνη τους. Έχουμε επίσης την έκθεση Μπρουκ που θα συζητηθεί αύριο το απόγευμα στην ημερήσια διάταξη ως προσθήκη. Συμφωνείτε μία δεύτερη μικρότερη αλλαγή σχετικά με την ημερήσια διάταξη. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής μας αύριο έχουμε μία μεικτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να ψηφίσουμε τους τρεις υποψηφίους ε, για το βραβείο Ζαχάροφ ε, που θα προτείνουμε στη διάσκεψη των Προέδρων και το έχουμε προβλέψει στις 5.30 ώρα. Λοιπόν, στις 5 όμως θα γίνει η συνεδρίαση, μισή ώρα νωρίτερα. Μπορούμε λοιπόν εμείς να δεχτούμε την ημερήσια διάταξη με αυτές τις αλλαγές, ωραία. Πάμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό θέμα. Έγκριση των πρακτικών της 1 η Σεπτεμβρίου. Τα έχετε στην, στα έγγραφά σας και αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα πρακτικά μπορείτε να ενημερώσετε τη γραμματεία πριν από το τέλος αυτής της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσεις της Προέδρου και θα τα πω αγγλικά γιατί οι σημειώσεις μου είναι στα αγγλικά. Δεν ε, θέλω να υποτιμήσω την γαλλική γλώσσα, απλώς η γραμματεία δεν ε, έχει τη δυνατότητα να συντάξει τις σημειώσεις στα γαλλικά. Η συνεδρίαση με τον ε, Ροζ Μιγκύρο θα διεξαχθεί στις, ε, τον 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Ενδεχομένω ε, να υπάρξει και μια έκτακτη συνεδρίαση την ΤΕΒΕ με την ΑΦΕΤ για τις εκλογές στο Αφγανιστάν και για τις επιπτώσεις τους ε, στο, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Γνωρίζετε ότι η εκλογέ στο Αφγανιστάν διεξήχθησαν στι 20 Αυγούστου. Τα αποτέλεσματα των εκλογών είναι κρίσιμη σημασία για το αφγανικό λαό και για την πολιτική σταθερότητα τη χώρα και για, το μέλλον, για το της περιοχής και τη ασφάλεια σε αυτήν. Γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει και τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, τον κύριο Καϊντ Άιντε, για μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ανάπτυξη και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των Αφγανικών εκλογών και περιμένουμε επιβεβαίωση πω θα έρθει να μα εντύσει στο Ασβούργο. Μόλι λοιπόν λάβουμε πληροφορίε, η Γραμματεία θα σα ανακοινώσει την ακριβή ώρα και τόπο τη συνεδριάσεω. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να μας ανακοινώσει κάτι. Νομίζω πως ο κύριος Γιάνσεν έχει κάτι να μας πει. Εγώ θα ήθελα να αναγγείλω στους, ε, στα μέλη ότι στις 17 ε, Σεπτεμβρίου η Κομισιόν ε, ενέκρινε την διετή της έκθεση για την ανάπτυξη η οποία διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο επαναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση στους 12 τομείς κλειδί. Θα υπάρχει δηλαδή μια συμβατότητα στις αναπτυξιακές, αναπτυξιακές πολιτικές, αναπτυσσόμενες χώρες. Και σας εύχομαι λοιπόν καλή ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις από την γραμματεία εγκαίρως. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται τρεις εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίασή μας. Περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της σχετικά με την συμμετοχή των μη κρατικών φορέων στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Οι μη κρατικοί φορείς είναι σημαντικοί εταίροι της Επιτροπής στην Ανάπτυξη, του 2007 περίπου 10% της ευρωπαϊκής, της ενίσχυσης της βοήθειας της Κομισιόν ε, έγινε από μη κρατικού φορεί. Έχουν οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια συγκριτικά πλέον εκτήματα κατά την υποστήριξη των τοπικών πληθυσμών μη κρατικοί φορείς λοιπόν και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνία των πολιτών ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία δημοκρατισμού των χωρών αυτών. Η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ανέκαθεν ε, θεώρησε ότι ο ρόλος αυτών των φορέων είναι πολύ σημαντικός κατά διάρκεια του δημοκρατικού ελέγχου και για την εφαρμογή της, του μέσου αναπτυξιακή συνεργασία η Επιτροπή συστηματικά του εάν όντως οι κοινωνίες των πολιτών συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην στη στρατηγική εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας. Έχουμε υποβάλει διάφορες ε, συστάσεις για να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Το Κοινοβούλιο επίσης υιοθέτησε και μια απόφαση για το έγγραφο της χρηματοδότησης αναπτυξιακής συνεργασίας. Τα έγγραφα αυτά θα τα βρείτε στο φάκελό σας. Σε ό,τι αφορά τώρα την παροχή βοήθεια στις χώρες ΑΚΕ, η Επιτροπή Ανάπτυξης σε τακτά διαστήματα έχει κάνει εκκλήσεις προς την Κομισιόν και θα πρέπει να διαπιστώσουμε το 2007 εν ώψη του 10 προγράμματος, ο πρώην Επίτροπος Λουί Μισελ ζήτησε από όλες τις ε, αντιμετωπίες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχουν σε αυτήν την συνεργασία. Επίσης ζητήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο να προετοιμάσει μια ειδική έκθεση για την ανάπτυξη και τη συμμετοχή συγγνώμη, των μη κρατικών φορέων στην συνεργασία για την ανάπτυξη. Αυτό το έγγραφο δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις αλλά και έχει και περιέχει συγκεκριμένε ε, συστάσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την ακρόαση σήμερα σε συνεργασία με την ε, Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν του συμμετέχοντες, τον κύριο Γιάνν Κίνστ, που είναι μέλο ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και εισηγητή τη ειδική έκθεση, την οποία συζητάμε σήμερα. Είμαι ευγνώμων που δέχτηκε την πρόσκλησή μα σήμερα και ε, παρατήρησα ότι είχε ήδη φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο για μια ανταλλαγή υποψίων με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ε, η δεσπενή κυρία Σιάν Πλάτ, η οποία είναι ε, σύμβουλος ε, της οργάνωσης World Vision. Σήμερα εκπροσωπεί το Concord που είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων για την βοήθεια και την ανάπτυξη. Το Concord εργάζεται στενά με τους εταίρους χώρες του Νότου και τον κύριο Κος Ρισελ, είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΑΕΤΚΟ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η DG ΑΕΤΚΟ συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής σε θέματα συνεργασίες με μη κυβερνητικούς φορείς. Μετά από την παρουσίαση θα ακούσουμε μια σύντομη παρουσίαση από τον συνάδελφό μας Μπαχστές που ως πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας είναι εισηγητής για την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κίνιστ που θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα και συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Κύριε Κίνιστ, έχετε το λόγο για 15 έως 20 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ακρόαση που μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα ευρήματα και πορίσματά μας. Η δική έκθεση ήδη συζητήθηκε νωρίτερα αυτό το χρόνο στο Συμβούλιο και στην Κόκομπή την περασμένη Πέμπτη. Χαίρομαι γιατί πολλοί εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται τόσο ζωηρά για την έκθεσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Στάις, τον εισηγητή της Κοκομπή, που έκανε τόσο ωραία σύνοψη της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό καταρχήν να διευκρινίσουμε τι είναι αυτή η μη κρατική φορείς, γιατί υπάρχουν πολλοί και διάφοροι ορισμοί στους κοινοτικού κανονισμούς. Συνήθως η έννοια μη κρατική φορείς καλύπτει όλες τις πτυχές της κοινωνίας που δεν αποτελούν κομμάτι του ιδιωτικού τομέα ή του κράτους. Συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπ' αυτή την έννοια χρησιμοποιείται και στην έκθεση το συνέδριο και το δικαστήριο χρησιμοποιεί τον ορισμό του κανονισμού που σε αντίθεση με την Συμφωνία του Κοτονού ε, δεν λαμβάνει υπόψη κερδοσκοπικούς φορείς. Επίσης υπάρχουν κοινοτικέ βάσεις, ε, ε, οργανισμοί, επαγγελματικοί, επιχειρηματικοί, περιβαλλοντικές ομάδες, ε, συνδικάτα, επιμελητήρια, εκκλησίες. Γνωρίζετε ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αναπτυξιακή συνεργασία ε, βάσει συνένεσης πέρασε από πολλές αλλαγές τα τελευταία δέκα χρόνια. Μεταξύ αυτών των αλλαγών η κοινοτική πολιτική όλο και περισσότερο θα συμπεριλάβει μη κρατικούς φορείς στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, αυτοί οι φορείς συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων που άμεσα ε, δίνουν ωφέλη για τους στόχους Η πολιτική της Ένωσης επίσης στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων ε, χιλίων περίπου μικρατικών φορέων για να παίξουν το ρόλο τους στο φως των παραπάνω και δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος πολλών εμπλεκομένων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συνέδριο αποφάσισε να κάνει έναν έλεγχο ούτως ώστε να κρίνει πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η συμβολή των μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον διπλό ε, ρόλο που έχουν ε, στην εταιρική, στις εταιρικές τους σχέσεις. Πρέπει να τονίσω ότι ήταν δύσκολο η ομάδα του ελέγχου να ε, παρακολουθήσει 100% τα οικονομικά αυτών των φορέων γιατί δεν υπήρχαν πολλά δεδομένα. Όμως Όλο και περισσότερο τα κονδύλια που δόθηκαν στους μη κρατικούς φορείς αυξήθηκαν την περασμένη δεκαετία και είναι το 10% περίπου πέρσι του, του γενικού προϋπολογισμού και ε, των, των αναπτυξιακών ταμείων και είναι περίπου 915 εκατομμύρια ευρώ. Το συνέδριο έθεσε τα εξή κέρια ερωτήματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει επαρκώ ότι οι μη κρατικοί φορεί συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία αναπτυξιακή συνεργασίας. Δεύτερον, το σύστημα διαχείρισης ε, της Κομισιόν διασφαλίζει ότι τα προγράμματα που εφαρμόζουν οι μη κρατικοί φορεί ε, πρόκειται να δώσουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, η Κομισιόν διασφαλίζει επαρκώς την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους μη κρατικούς φορείς. Θα ήθελα να συνοψίσω τα κύρια συμπεράσματα και συστάσεις με βάση το ελεγκτικό συνέδριο. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, διαπιστώθηκε ότι η Κομισιόν με τις αντιπροσωπείες της προσπάθησε να εντάξει τους μη κρατικούς φορείς στην προετοιμασία των στρατηγικών των χωρών σε όλες τις ε, δικαιούχους χώρες, της παραλήπτριες. Όμως η συμμετοχή ήταν ε, περιορισμένη, όπως σε, ένα, σε μια ημερίδα, ένα σεμινάριο μια ημέρα και δεν ήταν ο διάλογος αυτός ο δομημένος ο οποίος προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ειδικότερα το συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός για την διαχείριση και διευθέτηση όλων αυτών των διαδικασιών και υπήρχαν και καθυστερήσεις στη διανομή των εγγράφων. Επίσης υπήρχαν καθυστερισμένες ε, ε, προσκλήσεις ε, και ανεπαρκές feedback στους κρατικούς φορείς σε σχέση με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Αυτά τα πορίσματα είναι συνεπή με εκείνα της ίδιας της Κομισιόν. Δείχνουν ότι η μετάφραση των φιλόδοξων στόχων της ένταξης των μη κρατικών φορέων στις αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών σε πραγματικότητα παραμένει ακόμα μεγάλη πρόκληση. Όμως το συνέδριο αναγνωρίζει επίσης ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει και ε, καταλαβαίνει καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μη κρατικοί φορείς. Και οι δυσκολίες αυτές δεν ε, είναι φταίξιμο δικό τους, αναφέρονται. Επίσης ε, ε, ασχολήθηκε και με την ένταξη των μη κρατικών φορέων στην προετοιμασία θεματικών προγραμμάτων σχετικά με τις τοπικές αρχές και το ρόλο τους στην ανάπτυξη. Οι ε, ρυθμίσεις ε, και οι διαβουλεύσεις συμπεριέλαβαν χιλιάδε μη κρατικού φορείς, δεν οργανώθηκαν όμω αποτελεσματικά. Πάνω στη βάση αυτών των παρατηρήσεων συστήνει ότι οι Κομισιόν και οι υπηρεσίε τη θα πρέπει να δίνουν περισσότερε συμβουλέ προ ανατολισμό για το προσωπικό των αντιπροσωπιών, ούτω ώστε να ενταχθούν καλύτερα στην αναπτυξιακή διαδικασία οι μη κρατικοί φορείς, ε, προσφέροντα ε, εκπαίδευση κατάρτιση και ε, ενημερώνοντα τι κατευθυντήριε γραμμέ. Θα πρέπει επίση να εντοπιστούν σημαντική μη κρατική φορείς και να υπάρχει ένα πρόγραμμα διαβουλεύσεων. Θα πρέπει να επίσης να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι διαβουλεύσεων με τους μη κρατικούς φορείς σε κάθε χώρα χωριστά. Τώρα, η ε, διαχείριση, συστήματα διαχείρισης, ε, διαδικασίες επιλογής προγραμμάτων, έλεγχος, παρακολούθηση και διασφάλιση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων. Το συνέδριο διαπίστωσε ότι γενικά το σύστημα είναι στη θέση του ε, ώστε να επιλέγει τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα κατάλληλα προγράμματα ώστε να έχουν καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως ελλείψεις, ε, υπάρχουν θέματα ε, που μπορούμε να τα κρίνουμε θετικά σε σχέση με το θεμητό ανταγωνισμό, μπορούν όμως να υπάρξουν βελτιώσεις και για τις μη κρατικού και τις υπηρεσίες κομισιών. Η Κομισιόν πήρε μέτρα το 2006 και 2007 για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ε, προκήρυξης διαγωνισμού και μια διαδικασία επιλογής δύο βημάτων, όπου η πρώτη επιλογή θα στηρίζεται σε μια ε, σύντομη παρουσίαση με απερίληψη ε, των υπηρεσιών και μετά την πρόβλεψη ε, τοπικών ε, προγραμμάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, για διάφορα προγράμματα που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ανεπαρκής προετοιμασία, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμοστούν και αυτό επίσης ε, είχε αντίκτυπο στην, ε, για τον έλεγχο και την εποπτεία. Ε, αναγνωρίζει το συνέδριο τις προσπάθειες της Κομισιόν ώστε να εξοικειωθούν οι μη κρατικοί φορείς με το περιβάλλον των προγραμμάτων συμπεριλαμβάνοντας την ενίσχυση του διαλόγου με το Concord για θέματα συμβατικών υποχρεώσεων κλπ. και έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού και απλουστευμένες διαδικασίες και έντυπα. Όμως κάποιες ασυνέπειες στην ερμηνεία και την εφαρμογή των διαδικασιών καμιά φορά οδηγούσε σε άσκοπο διοικητικό φόρτο ε, σε βάρος των μη κρατικών φορέων. Επίσης επικρίναμε την ποιότητα του ελέγχου των προγραμμάτων που αξιολογήθηκαν από εξωτερικούς ελεγκτές. Και ε, τώρα θα πρέπει να να θεωρηθούν οι αρμοδιότητες ε, από το, και αυτό έγινε από το Φεβρουάριο του 2006. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται έλεγχος και παρακολούθηση το επίπεδο των ελέγχων ε, θα πρέπει να επεκτείνεται και στις συμβατικές υποχρεώσεις ε, υποστήριξη εγγράφων, ε, οι πολυπόμενες υποχρεώσεις, ε, συμπεριλαμβάνοντας και τα αναπτυξιακά προγράμματα των μη κρατικών φορέων. Επίσης διαπιστώνονται δυναμίες στον έλεγχο και την παρακολούθηση. Οι μηχανογραφημένες υπηρεσίες και συστήματα της Κομισιόν δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως. Τα δεδομένα είναι ατελή, και η αναγνώριση, ο εντοπισμό των υπεύθυνων δεν είναι αξιόπιστη και λίγες πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε ό,τι αφορά την ανάλυση και τη σύνθεση της κατάστασης των πραγμάτων ε, για τα συνεχιζόμενα και ολοκληρωμένα προγράμματα. Επίσης, ε, οι εκθέσει των έργων από τους κυβερνητικού φορείς που παίρνουν ε, δάνεια ή επιχορηγήσεις πολλές φορές δεν ε, συμπεριλαμβάνει καλή αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων, τίνοντας να υποβαθμίζοντας τις προβληματικές. Τέλος, ε, οι επισκέψεις που γίνονται από τις υπηρεσίες Κομισιόν είναι Έτσι λοιπόν συμφωνούμε με, σε αυτό το θέμα με τους μη κρατικούς φορείς ότι υπάρχουν ε, πολλά σφάλματα που μπορούν να αποφεύγονται αν βελτιώνεται η επικούρηση από την Κομισιόν. Ενώ τα προγράμματα που ελέγχθηκαν έχουν δώσει καλά αποτελέσματα ή βραχυπρόθεσμα θα τα δώσουν, οι προοπτικές για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους είναι περιορισμένα, κυρίως λόγω της μικρής διάρκειας του προγράμματος έργο. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μαζί με τις θεσμικές ρυθμίσεις που πρέπει να ε, βρεθούν είναι σημαντικές για την βιωσιμότητα. Πάνω στη βάση αυτών των παρατηρήσεων, το συνέδριο συστήνει η Κομισιό να συνεχίσει τα μέτρα ε, που ε, στοχεύουν στην βελτίωση της διαδικασίας δημοπράτησης και να φροντίζει ώστε η ε, τα έργα να κοινοποιούνται στους μη κρατικού φορείς και να υπάρχει αρκετή παρακολούθηση και υποστήριξη των αντιπροσωπιών και του προσωπικού των ε, μη κρατικών φορέων σε σχέση με δείκτες απόδοσης κλπ. Για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα, η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί μήπως πρέπει να ε, χρησιμοποιήσει ένα μίξ, ένα μείγμα ε, μέσων και όχι μόνο προγράμματα για τις, τους, μη, κρατικούς φορείς. Ο στόχος της ανάπτυξης ικανοτήτων σκοπό έχει να ενισχύσει το ρόλο των μη κρατικών φορέων και ως εταίρων στην αναπτυξιακή διαδικασία και ως φορέων υλοποίησης. Το συνέδριο σημείωσε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Προγράμματα για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κρατικών φορέων αναπτύσσονται και αποτελούν μέρος της ε, πρακτικής των περισσότερων χωρών και ενώ στις ασιατικές και λατινοαμερικανικές χώρες ε, δεν υπάρχουν ε, τέτοιες δυνατότητες, ε, ούτε προγράμματα. Αυτές οι διαφορές δεν προκύπτουν από μια συνολική αξιολόγηση αναγκών, αλλά αντικατοπτρίζουν απλά το γεγονός ότι η στήριξη, η ανάπτυξη ικανοτήτων ε, σε χώρες ΑΚΕ ήταν νομικό προ, προαπαιτούμενο στις χώρες ΑΚΕ, ενώ δεν ήταν στις ασιατικές και λατινοαμερικανικές χώρες. Επίσης, ο κανονισμός που ισχύει από το 2007 για τις ασιατικές και λατινοαμερικανικές χώρες προβλέπει ανάπτυξη ικανοτήτων για, τις, ε, για τους κυβερνητικούς φορείς, αλλά δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το πώς <clears throat> προσεγγίζεται το θέμα αυτό. Ο πρώτος γύρος των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων ήταν σημαντικός ε, στις παραλήπτριες δικαιούχους χώρες όμως ε, δεν έφτασαν, δεν το αξιοποίησαν 100% λόγω εγγενών περίπλοκων ε, διαδικασιών, συστημάτων και το εύρος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί και επίσης ε, ε, ε, δεν υπήρχαν ε, οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Επίσης είναι πολύ μακροσκελής οι διαδικασίες για την τεχνική υποστήριξη καταρχήν μετά για την προετοιμασία των ε, διαγωνισμών και τέλος αξιολόγηση προτάσεων και υπογραφή συμβάσεων, συμβασιοποίηση των έργων. Επίσης η δομή της διοίκησης με την κυβέρνηση, της, τους μη κρατικού φορείς, την αντιπροσωπείε της Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ε, είναι σαφής η ιδιοκτησία, αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο μέχρι να υπάρξει ομοφωνία. Η εφαρμογή των προγραμμάτων δεν ήταν πάντοτε επωφελής υπέρ αυτών που, των μη κρατικών φορέων που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη ε, την αναπτυξιακή. Ε, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν οι διαγωνισμοί για να επιλεγεί ο καλύτερος σε επιδόσεις μη κρατικός φορέας. Συχνά ε, κέρδιζαν οι αστικοί μη κρατικοί φορείς που είχαν καλύτερη χρηματοδότηση σε σχέση με τους άλλους στην Ήπεθρο με λιγότερα χρήματα. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων αυτών των φορέων στις ασιατικές και τις λατινοαμερικανικές χώρες και να γίνει μια διαφοροποίηση. Πρέπει να εξεταστούν πρόσθετοι τρόποι, ούτω ώστε να, ε, υπάρχουν, να ε, υπάρχουν οι στόχοι, να υλοποιηθούν δηλαδή, όπως εταιρικές σχέσεις, αμοιβαία χρηματοδότηση και προσπάθειες ώστε να φτάσουν στις, βάσεις, ε, στις οργανώσεις βάσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να ε, θίξω τα πιο σημαντικά συμπεράσματα ε, πορίσματα, συστάσεις. Υπάρχουν βεβαίως και πολλά άλλα πράγματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Τέλος, να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου προς τις υπηρεσίες της Κομισιόν για την καλή συνεργασία κατά, τον έλεγχο, κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Ελπίζω ότι η έκθεση από τον έλεγχο θα συμβάλλει σε μια πιο ενεργό συνεργασία των μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία των χωρών εκεί. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στη κυρία Πλάτ για 15 λεπτά. <laughs> I hope you will be able to see. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να προσθέσουμε και μερικές φωτογραφίες ε, στα λόγια μας, ε, διότι μερικές φορές ε, τα λόγια δεν επαρκούν και φαντάζομαι να λειτουργήσει το σύστημα. carry on. If technology defeats me, like civil society colleagues. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της τεχνολογίας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ που μας το καλέσατε σήμερα. Ονομάζομαι Σον Πλάτ και εργάζομαι για το Eurovision που είναι μια διεθνής ε, μη κυβερνητική οργάνωση και προσωπεί το δίκτυο Concord. In case you're not familiar, Concord is the European NGO Confederation for Relief and Development. Η οργάνωσή μου έχει πάνω από χίλιες, πάνω από χίλιες οργανώσεις που δουλεύουν σε διάφορες πλατφόρμες και προσωπούν χιλιάδες ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, που δείχνουν ενδιαφέρον ανάπτυξης ε, και βοήθειας τόσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά όσο και σε επιτόπια δράση. Η Concord έχει σημαντική διάδραση με αυτές τις επιτροπές και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ένα ιδιαίτερο επικοδομητικό διάλογο. Θα προσπαθήσω να παραμείνω μέσα στα χρονικά όρια αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο με τους ε, ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, ποια ήταν η αντίδρασή μα στην έκθεση. Θα θέλουμε να πούμε, συμφωνούμε με το ελεκτικό συνέδριο, αλλά φυσικά έχουμε κάποιες περισσότερες ε, περισσότερες ε, ιδέες πάνω στο θέμα και προσδοκίες. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πραγματικότητα που επικρατεί στις διάφορες οργανώσεις αλλά και στους ντόπιους πληθυσμούς. Υπήρχε ένα σεμινάριο στο Παρίσι το, 2004 όπου η Κοκόρτ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν τα μέσα για την πρόθεση του διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκομένους και κάναμε κάποιες συστάσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και κοιτάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται. Υπάρχει λοιπόν η βούληση να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη. Πρώτο σημείο. Το συνέδριο έφυξε το ζήτημα της συνεργασίας και του διαλόγου. Ξέρετε ότι ο διάλογος δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί και χρειάζεται πολιτική βούληση αλλά και εφαρμογή αυτού. Αυτής, ε, αυτό απαιτεί αλλαγές ε, σε κάποια όργανα σε ό,τι αφορά την νοοτροπία, κάτι το οποίο έχει προτεραιότητα πριν να ε, περάσουμε στο επίπεδο διαχείρισης πολύ συχνά διαδικασίες και η χορήγηση πόρων καθορίζονται από την ανάγκη να ελεγχιστοποιηθεί ο χρόνος και για πιο άμεση χρηματοδότηση. Φαίνεται ότι η Κομισιόν βρίσκεται πιο εύκολο να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς ε, όπως η Vision από τη μικρή οργανισμή γιατί έτσι καμιά φορά εκπληρώνουν αποτελεσματικότερε στόχε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Κομισιόν χρειάζεται να βρει περισσότερη βοήθεια από τι ε, οργανώσει οι οποίε δρούν επί τόπου. Εδώ και καιρό ε, το που συνεργάζεται με το EuroPaid προκειμένου να βελτιωθούν αυτοί οι μηχανισμοί όπως ο δημοσιονομικός κανονισμός και Υπάρχει γενική συνένεση ε, στην Ευρώπη ανάμεσα στους θεσμούς για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. στο σύνοδο του των Παρισιών, του των Παρισίων, εξετάσαμε αυτό το ζήτημα και καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία να ε, είναι αποτελεσματικότερη και να υπάρξει συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Θα σα δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες. Ε, βλέπετε τώρα έναν άνθρωπο σε ένα κουτί. Ε, υπάρχει μια λιγορία εδώ. Και αφορά στη συνεργασία μας με το πλαίσιο που μας, που Δεν ε, μας αρέσει και πολύ αυτός ο κύριος ο οποίος στριμώχνεται μέσα στο κουτί. Και το ελεγκτικό συνέδριο έχει εντοπίσει τι ε, δυσκολίε που υπάρχουν ε, σχετικά με την βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τώρα μικρά παραδείγματα, όπως τα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να μπούμε λοιπόν μέσα σε, κάποιες, σε κάποια χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να τηρηθούν είναι δύσκολο να συμμετάχουν σε μια συνεργασία όταν έχει κανεί δύο μέρε μόνο να μεταβεί σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε μια χώρα τέσσερι φορέ μεγαλύτερη από το Βέλγιο και με πολύ χαμηλέ υποδομέ. Το ζήτημα του χρόνου λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για τι ε, οργανώσει ε, αυτέ, ε, οι οποίε δεν έχουν πάει την δεν έχουν απόλυτη ευελιξία. Χρειάζεται λοιπόν πολλές φορές ε, να βρούμε, να είμαστε κάπως πιο εφάνταστοι για να προωθήσουμε τα προγράμματά μας. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε περιορισμούς και να μπαίνουμε μέσα σε ένα μανδύα. Θα προτιμούσαμε λοιπόν να υπάρξει μια εταιρική σχέση η οποία θα μας επιτρέψει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και να περπατάμε λίγο πιο άνετοι. Τώρα υπάρχουν ε, κάποια κενά στην πολιτική. Η συνεδρίαση των δωρητών στην Άκρα ε, έδειξε ότι οι δωρήτριες χώρες ε, μερικές φορές ε, δεν καταφέρνουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την κοινωνία των πολιτών. Πάντως, μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών απουσιάζει μια κοινωνία των πολιτών που θα μπορούσε να βασιστεί σε μια πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία. Έλλειψη λοιπόν προγραμμάτων και κατάλληλης ε, χρηματικής στήριξης είναι κάτι το οποίο αναφέρει και το ελληνικό συνέδριο. Το χρηματοδοτικό μέσο μερικές φορές δεν καθίζει τόσο αποτελεσματικό διότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός και σε γεωγραφικά προγράμματα όπως το EDF υπάρχει πρόβλημα υποχρηματοδότησης ε, για κάποιες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και το Κονκόρντο όπως και το συνέδριο φρόντισε να, δείξει, να καταδείξει την έλλειψη διαφάνειας ε, που υπάρχει. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά στο μέλλον και οι ε, υπάρχουσες πόροι του, του συστήματος θα πρέπει να έχουν καλύτερη εκμετάλλευση. Εμείς ε, συμφωνούμε με κάποιες προτάσεις του συνεδρίου, αλλά η ε, Concord θεωρεί ότι ε, πολλά από τα κονδύλια δεν μπόρεσαν να, να δαπανηθούν ακόμα, κάτι το οποίο σημαίνει μια έλλειψη αυτών αποτελεσμάτων. Οι συζητήσεις που είχαμε με άλλου ενδιαφερομένου, διότι η Concord αποτελεί ένα κομμάτι τη κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις λοιπόν των πολιτών, παρατηρούν ότι το, οι κανονισμοί μερικέ φορέ είναι δυσκίνητοι και το άχθος το οποίο προκαλούν είναι ιδιαίτερα βαρύ. Θα κάνω αυτή την παρουσίαση λίγο στα, στα βιαστικά, διότι δεν έχω αρκετό χρόνο στη θέση μου. Το ε, θέμα της ε, λογοδοσίας είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τις κοινωνίες των πολιτών στο θέμα της ε, λογοδοσίας και απέναντι στις ε, οργανώσεις που δουλεύουν αλλά και απέναντι στους δωρητές. Υπάρχει λοιπόν πολύ σημαντικό να, είμαστε, υπάρχει λογοδοσία απέναντι στους ε, δωρητές. Δεύτερον, αξιολογώντας την εργασία της κοινωνίας των πολιτών και τον ορισμό νέου προγραμμάτων θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Συμφωνούμε με το Ελληνικό συνέδριο πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, βιωσιμότητα των προγραμμάτων. επίση τονίζουμε ότι πολλέ αξιολογήσει κατέδειξαν ότι η συνεργασία ανάμεσα στι ε, οργανώσει μπορεί να διασφαλίσει την βιωσιμότητα. Τρίτον, ε, να μην να φροντίσουν να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων για την απόκτηση πόρων η δυναμική έχει αρχίσει να αλλάζει και αυτό το έχουμε καταγράψει. Αλλά το να έρθουμε σε αντίθεση, να έρχονται σε αντίθεση οι οργανώσει μεταξύ τους είναι κάτι το αντιπαρογικό. Δεύτερον, να υπάρξει συμμετοχή των Κοινωνία των πολιτών σε προγράμματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον διάλογο. Πιστεύουμε πως ε, αν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα έχουμε μια απώλεια της ευκαιρίας, χάσουμε τις ευκαιρίες που μας ε, προσφέρονται. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια συνεργασία από την κορφή προς τη βάση και τούμπαλιν. Ε, πέμπτο, να υπάρχει συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών με τις ε, τοπικές αρχές. Οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών έχουν μακρά ιστορία σε συνεργασία, θέματα συνεργασία με, το με το αυτοδιοίκηση. Αυτό βελτιώνει την διακυβέρνηση και καθιστά υπόλογου ε, του ε, υπολογιστή οργανώσει. Έκτον, ε, έχουμε να δημιουργήσουμε απαραίτητους να διέσουμε του απαραίτητου πόρου έτσι ώστε να γίνει πιο ενεργή η κοινωνία των πολιτών. Όλες οι κυβερνήσεις ε, υποστηρίζουν τις οργανώσεις αυτές Δεύτερον, να αναζητήσουμε ελληνικές μέθοδους για τη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, συγγνώμη, τις κοινωνίες των πολιτών. Το ισχύοντα σύστημα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Αυτό φυσικά θα βελτιώσει την ε, αποτελεσματικότητα των πόρων. Χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια, Όγδον, να υποστηρίξουμε τις ε, πρωτοβουλίες ε, της κοινωνίας των πολιτών. Ελπίζω να γνωρίζετε τις ε, πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτελεσματικότητας. Εάν δεν το γνωρίζετε, παρακαλώ ενημερωθείτε σχετικά. Οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, ε, απανταχού όχι μόνο στην Ευρώπη, προσπαθούν να προσδιορίσουν τι σημαίνει αποτελεσματικότητα και έχουν εντοπίσει τι βέλτιστε πρακτικέ που υπάρχουν σε ζητήματα λογοδοσία. Ίσως να αισθανθείτε όπω ε, οι χαρακτήρε σε αυτό την ε, γελιογραφία που δείχνουν τι διάφορε τάσει που υπάρχουν χρηματοδότηση. Τώρα, προς τα που πηγαίνουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία επισημαίνει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η Concord είναι μέρος της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της. Ήδη έχουμε κινητοποιήσει ιδέες και πόρους για να ανταποκριθούμε σε κάποιες από τις συστάσεις. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε πως η σημασία αυτού του διαλόγου ε, τη χάνει εκμετάλλευση ε, ε από όλους τους εμπλεκομένους και οι οποίοι συμμετέχουν στις ε, συζητήσεις ε, το Κοινοβούλιο θα είναι ένα βασικός παίκτη ε, και θα θέλαμε να συζητήσουμε και με την Επιτροπή και με Επιτροπές του και τώρα για τις μελλοντικές εξελίξεις πρέπει να αξιολογήσουμε, να διασφαλίσουμε την συνεργασία προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ε, ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων και να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Μια σοβαρή έκθεση απαιτεί σοβαρή απάντηση. Η έκθεση του συνεδρίου αναλύει την κατάσταση και απαιτεί δράση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια. Το G20 αναγνώρισε την σημασία της ε, εξάλληψης ε, της ε, φτώχειας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μπορέσουν οι μη κυβερνικές οργανώσεις να δερματίσουν τον ρόλο τους. Πιστεύουμε λοιπόν πως ε, μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Mr. you have the floor for... Ο κύριος Ρισέλα έχει το λόγο από την Κομισιόν για να απαντήσει στις επικρίσεις, ερωτήσεις, θέσεις για 15 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα 15 λεπτά όπως μου είπατε. Είναι πολλά για να αντιδράσω στα όσα ακούσαμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα αρκέσουν. Εγώ πάντως θα τα τηρήσω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας επέτρεψε να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις αυτές επί της πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου που χαιρετίζομαι και που στις αντιδράσεις μας ε, δείχνουμε πόσο την εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πολύ και από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, το έγγραφο εργασίας του κυρίου Στάζ, τα συμπεράσματά του είναι νομίζω πάρα πολύ καλά ισορροπημένα. Η κυρία Πλάτ τελείωσε την έκκλησή της λέγοντάς, ότι, λέγοντάς μας ότι μια σοβαρή έκθεση απαιτεί σοβαρή απάντηση, αντίδραση. Αλλά δεν μπορεί να είναι η αντίδραση αυτή μόνο της Κομισιόν. Είναι πολύ οι στον τομέα αυτό. Όχι μόνο οι μη κρατικοί φορείς, αλλά οργανώσεις, ιδρύματα, θεσμοί, όπως ε, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια πολιτική, μας βρίσκει σύμφωνος ε, η σημασία των μη κρατικών φορέων, κανείς δεν αμφισβητεί, κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει τη σημασία του στην Κομισιόν και όλοι θέλουμε να την ε, πραγματοποιήσουμε την πολιτική. Η διαφορά τώρα μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να συντρέχουν όπως νομοθεσία και ε, συγκεκριμένα εμπόδια που πρέπει να υπερκεραστούν, υπερπηδηθούν και στοιχεία βέβαια. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τι ε, παίρνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γνωρίζουμε όμως, υπολογίζουμε ότι περίπου είναι το 10%. Δηλαδή ένα δις ετησίως δαπανάτε με αυτόν τον τρόπο και σε αυτούς τους φορείς. Πολλά πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία και σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Αυτά όλα θα πρέπει να ανακαινιστούν, να έχουμε καινοτόμες καινούριε μορφές συνεργασίας. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο με τη ρυθμό απόδοση, τις εισρωές, πρέπει να έχουμε και την απόδοση υπόψη μας, δηλαδή τα αποτελέσματα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε την υποδομή, τις προσλαμβάνουσες της κάθε χώρας, ε, ε, τη, την νοοτροπία που υπάρχει και θα πρέπει ανάλογα να προσαρμόσουμε το πώς κινούμεθα. Παλιότερα, ε, προηγουμένω ε, στην Επιτροπή Κοκομπή, κάναμε ενδιαφέρουσε συζητήσει για τον ορισμό του μη της μη κυβερνητική οργάνωσης. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια οργάνωση που επιδοτείται 100% από δυο κυβερνήσεις ή την Κομισιόν και μια κυβέρνηση ή θα πρέπει να έχουν τα δικά τους τα χρήματα, ε, το δικό τους χώρο που πρέπει να καλύπτουν, να έχουν δηλαδή μια περιφέρεια που να καλύπτουν. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και ποια θα είναι η συνεργασία τους με τους μη κρατικούς φορείς ε, γενικότερα. Ε, αποτελεσματικός διάλογος ε, ετέθη αυτό το θέμα με χώρες εταίρους ή με εταίρους γενικότερα. Αν το καταπιαστούμε αυτό το θέμα, αμέσως ε, μπαίνει το θέμα της ιδιοκτησίας ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που έχουμε, αυτό είναι απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να το οργανώσουν έτσι, είναι οι γεωγραφικοί προϋπολογισμοί. Και επί αυτής της βάσεως συζητήσαμε με τις κυβερνήσεις των αποδεκτριών, αποδεκτριών παραληπτηριών χωρών. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε περισσότερους μη κρατικούς φορείς σε αυτή τη διαδικασία αλλά θα πρέπει να ε, κάνουμε έκκληση, να, να τους πείσουμε, δεν μπορούμε να τους ε, αναγκάσουμε. Πρώτα θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με την κυβέρνηση της ε, δικαιούχου χώρας και μετά να πάμε στην στο μη κρατικό φορέα. Η καλή συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αφορά και τα κοινοβούλια, που πολλές φορές δεν συμμετέχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες στην κατάρτιση τέτοιου είδους, τέτοιου είδους προγραμμάτων, σχεδίων κλπ. Μην κάνετε λοιπόν το λάθος και πείτε ότι δεν επιμένουμε εμείς και δεν πιέζουμε. Βεβαίως και πιέζουμε ώστε να συμμετέχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά σε τελευταία ανάλυση υπάρχει και μια πραγματικότητα επί τόπου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, ακούσαμε παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας, των δράσεών μας, σε ό,τι αφορά την ένταξη ε, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων στην δημιουργία ικανοτήτων. Εδώ είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ένας ολόκληρος κόσμος. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Τώρα έχουμε ένα σύστημα αυτοεγγραφής ε, ε, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και έχουμε πολλές χιλιάδες. Αν λάβουμε υπόψη μας την ε, δημιουργία ικανοτήτων και μιλάμε και για περίπου 15.000 εγγεγραμμένες οργανώσεις με μεγαλύτερο δυναμικό, πώς θα τους οργανώσουμε αυτούς τους φορείς και πώς θα τους οργανώσουμε μάλιστα και με βιώσιμο τρόπο γιατί υπάρχουν αλλαγές στην ηγεσία, στο ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την, τον ηγετικό ρόλο. Και αυτά δεν είναι μέρος της περιγραφής των ε, ε, δραστηριοτήτων μας. Δεν είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και από την άλλη υπάρχει και περιορισμός του τι μπορεί κανείς να κάνει σε μια χώρα. Οργανώνουμε ενημερωτικέ εκδηλώσεις, ε, προβαλόμεθα από το website, έχουμε ε, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, αλλά αυτά δεν ακούν για να φτάσουμε ούτε και σε ένα μεγάλο ποσοστό των 15.000 οργανώσεων. Υπάρχει όμως η δυνατότητα γιατί αν θέλετε είναι ένα όνειρο αυτό το ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες για όλους. Τώρα, η βιωσιμότητα. Ε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας. Υπάρχουν ε, ολόκληρες βιβλιοθήκες θέλω εγώ, ε, που περιλαμβάνουν προγράμματα βιωσιμότητας και μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχολείο ας πούμε, να το ετοιμάσουμε, αν όμως μετά το Υπουργείο γυρίσει την πλάτη, τότε ποιος θα πληρώνει τους μισθούς των εκπαιδευτικών, ποιος θα προμηθεύεται τα βιβλία. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια βιωσιμότητα καταβολή μισθών κλπ. Αυτά τα λέμε και στη, στα έγγραφα πολιτικής μας. Και υπ' αυτή την έννοια ε, κάνουμε τομεακή υποστήριξη και ε, υποστήριξη του γενικού προϋπολογισμού. Δεν αποκλείουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά μια φάση αργότερα. η κυβέρνηση της χώρας εταίρου ε, θα ε, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων επικουρούμενη και από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους μας. Έχουμε κάνει μια ανοιχτή συζήτηση και με το Concord και με άλλες οργανώσεις, αλλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε, τι εννοούμε, και πώς μπορεί να ενταχθεί και στον, ε, στην ανάπτυξη των τομέων η κοινωνία των πολιτών και στην υποστήριξη του προϋπολογισμού. Στα πλαίσια της βιωσιμότητας είναι επίσης πολύ σημαντικό να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στην χαρτογράφηση, αν θέλετε, των τεκτενομένων σε μία χώρα και από την κοινωνία των πολιτών και τους επίσημους δωρητές. Και να ξέρει η δεξιά τύπη η αριστερά να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί πώς συντονίζονται. Ε, και βεβαίως να ξέρουν και τι κάνει η κυβέρνηση μιας δεδομένης χώρας για να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους ε, δρόντες που παρουσιάζονται επί τόπου. Τώρα για τις διαδικασίες μας, μάλιστα είναι ε, επίπονες, έχουμε κάνει συγκρίσεις και με άλλους δωρητές και φαίνεται ότι από την αρχή των προγραμμάτων μέχρι την πρώτη απόφαση δεν είμαστε πιο πίπονοι στις διαδικασίες, δεν έχουμε πιο επαχθείς διαδικασίες από ότι οι ε, αγγλικές, οι γαλλικές ε, ε, οργανώσεις. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που παίρνουν χρόνο. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι εμείς θα και είμαστε πιο χρονοβόροι. Είναι πολύ τεχνικές διαδικασίες που αντικατοπτρίζονται σε ένα δημοσιονομικό κανονισμό αποδεκτό από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Την περασμένη φορά κάναμε μια απλούστευση και κάναμε 150 προτάσεις απλουστευτικές. Μόνο 25-26 από αυτές επιβίωσαν τις διαδικασίες δηλαδή που πέρασαν από τα διάφορα στάδια των διαπραγματεύσεων. Και πάλι θα υποβάλλομαι ε, καμιά ε, 115 περίπου θα κάνουμε απλουστευτικές προτάσεις για τον, να απλουστεύσουμε τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και θα δούμε τι θα γίνει. Έχει, εφαρμόζεται, αλλά υπάρχει ένας κανονισμός που λέει στο άρθρο 42 ότι είναι κανείς υπεύθυνος για σοβαρά λάθη. Αυτό δεν είναι ο, η καλύτερη ενθάρρυνση για να αναλάβει κάποιος και ένα ρίσκο. Από τη μια ζητούμε από την κοινωνία των πολιτών να αναλαμβάνει περισσότερο ρίσκο και από την άλλη έχουμε τους ελεγκτές ε, του συνεδρίου του ελεγκτικού που ε, φρενάρουν. Ε, βέβαια, λένε να προσέχουν πολύ. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ στα σημεία που εκπέμπουμε και θα πρέπει να τα συγκεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, αλλά δεν είναι δυνατόν να κινηθούμε στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού προς μια συγκεκριμένη ρύθμιση διακανονισμό όπου μια ομάδα ε, φορέων θα ε, επιλεγούν και θα πούμε αυτή είναι η καλύτεροι, με αυτού θα δουλεύουμε. Όχι. Πάντα θα πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί που παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και αναπόφευκτα οδηγούν σε απογοήτευση των δύο τρίτων των ανθρώπων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, γιατί ο προπολογισμό είναι πεπερασμένο και δεν μπορούμε να δεχτούμε πολλέ προτάσει. Πάντα με ενδιαφέρει να, ε, να ακούω ότι εφαρμόζονται καινοτόμιμες μέθοδοι και προσπαθούμε να δούμε, ας πούμε, να έχουμε τέτοιες μικρές σφήνες καινοτόμου, Ήδη είμαστε στη διαδικασία της προετοιμασίας των ε, προτάσεων για την απλούστευση, απλοποίηση που θα πρέπει να συζητηθεί για το 2010. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, για τη διαδικασία του Παλέρμο, αυτός ο τετραμερής διάλογος που οργανώσαμε από το 2003 ε, τώρα θα αποσταλεί και νέα πρόσκληση για να αναζωογονηθεί ο διάλογος και να καθίσουμε τέλος πάντων με τους τέσσερις εμπλεκομένους στη συζήτηση αυτή και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να συνεχίσουμε. Αν αποκομίσατε την εντύπωση ότι η παρέμβασή μου ήταν αμυντική, σφάλετε. Εγώ έθεσα επιτάπητος ορισμένα θέματα τα οποία τα βλέπουμε και στην πράξη να εμφανίζονται και έχουν σχέση με την πρακτική δυσκολία της πρακτικής εφαρμογής, της εφαρμογής στην πράξη των κανονισμών και των οδηγιών. Όμως ε, τα χρήματα δαπανώνται, αυτό που αναμένεται από μας το παραδίδομαι και πάντοτε υπάρχει τρόπος για να λειτουργούν τα πράγματα. Πολλές φορές ανεβαίνει η αδρεναλίνη και πολλές φορές κανείς θαυμάζει και λέει είναι θαύμα πώ μπορέσαμε να δαπανίσουμε με καλό τρόπο τα χρήματα που έχουν διατεθεί. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα και τους επόμενους μήνες θα πάμε ακόμα καλύτερα γιατί θα ε, απλουστεύσουμε, θα προτείνουμε να απλουστευτεί περισσότερο ο δημοσιονομικός κανονισμός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρισελ. Ο κύριος Μπαρτ Στάις έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι απόλυτα λογικό στην Κατά την επόμενη θητεία, μάλλον σε αυτήν τη θητεία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ αυτής της Επιτροπής και του ελέγχου προϋπολογισμού. Στο παρελθόν υπήρξε μια ε, αξιοθρύνητη σχέση μεταξύ μας. Εγώ σε αυτήν την Επιτροπή είμαι αναπληρωματικός, αλλά στον έλεγχο του προϋπολογισμού Είμαι πρώτος αντιπρόεδρος και δεσμεύομαι στο μέλλον η συνεργασία να είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι στο παρελθόν με μια γρήγορη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Μετά από αυτά να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο στο παρελθόν ε, συνέταξε εκθέσεις για τη συνεργασία ε, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Έχουμε μία έκθεση για την τεχνική βοήθεια, για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού τον Μάρτιο και τον Απρίλιο της ε, ε, προηγούμενης θητείας. Έχουμε επίσης μία έκθεση για την υγειονομική βοήθεια στην υποσαχάρια περιοχή. Και όλα αυτά κατέληξαν σε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μας υποστήριξε και έλαβε υπόψη της τα αιτήματά μας. Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε κάτι το συγκεκριμένο και θετικό. Τώρα, μετά την ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την εργασία, διότι πρόκειται για μια έκθεση πάρα πολύ συγκεκριμένη ε, και λεπτομερή. Και σε αυτή την έκθεση γίνονται μερικές, ε, δίνονται μερικές διατυπώσεις ε, σαφέστατες, ε, διότι το, το ελεγκτικό συνέδριο δεν διστάζει να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για μας ε, για να μπορέσουμε να, ε, να ξεκινήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Μετά λοιπόν από την ανάγνωση της έκθεσης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος ε, Ρισελ ε, μας είπε ότι η τοποθέτησή του μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αμυντική σήμερα. Εγώ δεν είχα καμία τέτοια αίσθηση ακούγοντας τον εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σωστή αντιμετώπιση, διότι υπάρχουν ένα σωρό αιτήματα διότι ε, είχαμε την τελευταία διετία της προηγούμενης ε, θητείας 4.500 ε, αιτήματα για ενίσχυση της τάξης των 280 ευρώ και μόνο το 4,6% των διαφόρων αιτημάτων που διατυπώνονται μπορούν να καλυφθούν Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια πρόκληση όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Επίσης υπάρχουν τεράστιοι περιορισμοί που μας επιβάλλονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό και πρέπει να τον ε, σεβαστούμε. Διότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζεται από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστός. Υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες σίγουρα θα πρέπει να έρθουν Οι υπάλληλοι που πρέπει να αποφασίσουν είναι οι υπεύθυνοι για αυτές ε, τις αποφάσεις. Δεσμεύονται, έχουν την ευθύνη, δεσμεύοντας την ίδια τους την περιουσία ε, πρέπει να έχουμε λοιπόν επίγνωση όταν λαμβάνουμε οικονομικές αποφάσεις και πρέπει να σεβόμαστε συνεχώς ε, όλα όσα μας ε, αναφέρουν όσοι εργάζονται επί τόπου. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο η οποία λέει ότι η Κομισιόν ε, υποβάλλει πάρα πολύ καλές προτάσεις ε, και θέλει να υλοποιήσει το αναπτυξιακό, το αναπτυξιακό όνειρο, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω των τεραστίων διαφορών ε, των καταστάσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταγράφηκαν και οι 15.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε έναν κατάλογο, οι οργανώσεις που εργάζονται σε αυτές, ε, σε αυτές τις ε, περιοχές ε, για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι ιδιομορφίες της κάθε περιοχής. Τώρα, εγώ ως εισηγητής για την απαλλαγή θεώρησα ότι πρέπει να λάβω υπόψη μου τέσσερις με πέντε ε, συστάσεις για την έκθεση που θα κατατεθεί στα, τον Νοέμβριο και με τον κύριο Λιμπεράσκη, α, σοσιαλδημοκράτη εισηγητή, είπαμε να δούμε ξανά τις αντιπροσωπίες και να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα άτομο από κάθε αντιπροσωπεία το οποίο όχι μόνο να έχει υπόψη του το πώς λειτουργεί η δημοσιονομική διαδικασία αλλά να ε, είναι γνώστης για το τι γίνεται επί τόπου, διότι επί τόπου αντιμετωπίζονται όλες οι προκλήσεις. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν γνώση της κάθε κοινωνίας των πολιτών και της κάθε ιδιάζουσας κατάστασης για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. η Κομισιόν έχει σίγουρα δυσκολίες για, το, για τη χορήγηση αυτού του δισεκατομμυρίου ε, σε, σε μικροπιστώσεις. Αλλά εν ώψη της έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2011 δεν θα έπρεπε όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας ακριβέστερα δεδομένα από την Κομισιόν να εγκρίνουμε τη χορήγηση πιστώσεων σε όσο το δυνατόν πιο μικρές μονάδες της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, η αναπτυξιακή πολιτική σε αυτό το κοινοβούλιο καλύπτεται από την αρμοδιότητα πολλών επιτροπών. Και αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε το όλο σύστημα χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών ώστε να υπάρχει διαφάνεια και παραγωγικότητα στις ε, διαδικασίες μας, ώστε οι πολίτες ε, να μπορούν να βασίζονται στην, στην πολιτική μας αυτή. Επίσης, ζητείτε και μία αξιολόγηση της όλης διαδικασίας του Παλέρμο. Έχουμε φτάσει τώρα στην ε, φάση του Παλέρμο 2. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε έναν απολογισμό. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό, ώστε οι προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν να αποτελέσουν τη βάση των διαβουλεύσεων για αυτόν τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης έχει λάβει υπόψη της <coughs> διάφορες συστάσεις αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες από την ε, Κομισιόν για την ε, προώθηση και της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει λοιπόν να τις λάβουμε όλες υπόψη μας. Τον Απρίλιο του χρόνου θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της απαλλαγής για το 2008. Λοιπόν, είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής και είμαι έτοιμος να εργαστώ γι' αυτό. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ε, ερωτήσεις ε, και παρακαλώ μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ε, στους εμπειρογνώμονες. Ο κ. Βέραν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Εύα Ζολή. Κατά την άποψή μου, η έκθεση αυτή χρειάζεται μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση. Θεωρώ πως ε, αυτή η κριτική που ασκείται στην έκθεση είναι τόσο εντυπωσιακή και θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε κάποιες περαιτέρω προφορέ από την Ευρωπαϊκή Τροπή. Πολύ μετριοπαθής ήταν η αντίδραση. Φυσικά όλοι κατανοούμε τις δυσκολίες ε, που υπάρχουν στον τομέα. Όταν κανείς εργάζεται με 15.000 οργανώσεις μη κυβερνητικέ, είναι κάτι το πολύ περιπλόκο. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να κάνουν το δικό τους ε, κομμάτι δουλειάς και να υπάρχει καλύτερο συντονισμό από αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά δεν αφορά αυτό μόνο τις μη οργανώσεις. Αφορά και την προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που θα πρέπει να καταδείξουν ότι το ζήτημα απαιτεί μια νέα προσέγγιση στο θέμα της συνεργασίας ε, με μη κρατικές οργανώσεις Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ε, τόσο ημών όσο και των ε, οργανώσεων. Τώρα, εάν ε, οι κατοχώρες έχουν κάποιες επιτυχίες στο Αφγανιστάν, αυτό οφείλεται μόνο και μόνο στο ότι η αναπτυξιακή πολιτική των κάτω βασίζεται σε μια σχέση κατάντη ανάντη, δηλαδή στην στενή συνεργασία με τους επιτόπου φορείς. Κάτι το οποίο δεν κατανόησαν ποτέ οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν, αλλά και αλλού στον κόσμο. Λοιπόν, τι πρόκειται να πράξει η Ευρωπαϊκή Ευρωπή σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε. Δεν άκουσα λοιπόν από τον κύριο Ρουσέλ τι προγραμματίζει να πράξει κατανοώ πως υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της ε, επένδυσης σε ζητήματα ανάπτυξης ικανοτήτων, διότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανταπόκριση, μια αντιστοιχία ανάμεσα στην κονδύλια τα οποία χορηγεί κανείς για την ανάπτυξη ικανοτήτων και το αποτέλεσμα που αποφέρουν. ως Ευρωκοινοβούλιο πιστεύω πως ε, πρέπει να έχουμε μαζί μας ε, αυτή την έκθεση όταν ασχολούμεθα με θέματα δημοκρατικού ελέγχου, ανεπεξιακής πολιτικής κλπ. και να αναρωτιόμαστε πάντο πόσο σημαντική και αποτελεσματική είναι η συνεργασία κομισιών ε, με κυβερνητικών οργανώσεων σε ένα χρόνο θα πρέπει να δούμε τι θα έχει αλλάξει στην προσέγγιση της Κομισιόν σχετικά με την ε, συμμετοχή και ανάμειξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ανάπτυξη βοήθεια. Αυτά ευχαριστώ. Merci. Je donne la parole à Monsieur Ευχαριστώ, κύριος Γκερέρο, έχει το Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και, στο, και το ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εμπειρογνώμη μας κυρία Πλάτ για τις παρουσιάσεις μας έκαναν και κανείς δεν αφισβητεί σήμερα τη σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, εργασίες κλπ που το καταδεικνύουν αυτό, αλλά επίση υπάρχουν και πάρα πολλές ε, πολιτικές ε, εντολές θα έλεγα. Ε, η κυρία Πλάτα αναφέρθηκε σε τρεις εξ αυτών. Η ατζέντα της Άκρα, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της Αφρικής. Δεν αφισβητείται λοιπόν πως η πολιτική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει μια βάση ε, αποτελεσματική. Τώρα, το ελεγκτικό συνέδριο αυτό το οποίο δηλώνει είναι πως ε, βρισκόμεθα ενώπιον περιορισμών προκειμένου να υπάρξει πλήρη συμμετοχή των μη κρατικών φορέων. Οι περιορισμοί είναι γεωγραφικού χαρακτήρα αφενός, λειτουργούν στις χώρες ΑΚΕ, αλλά δεν λειτουργούν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η Λατινική Αμερική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ανεξιακής μας πολιτικής. Επίσης υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά τους εμπλεκομένους. Στην ανάλυση του Συμβουλίου αναγνωρίζεται ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε, να ανοιχθούμε μάλλον σε περαιτέρω μη κυβερνητικούς, μη κρατικούς φορείς. Και επίσης υπάρχουν και περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις ικανότητες των μη κρατικών φορέων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προτείνουμε εδώ μία περαιτέρω ενημέρωση και αυτών των ε, μη κρατικών ε, φορέων. Εδώ έχουμε τρεις στόχους που θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Δεύτερο, πρώτον, να διευρυνθεί εδαφικά θα λέγαμε η συμμετοχή των μη κρατικών φορέων, να διευρύνουμε περαιτέρω τον αριθμό τους και να τους καταρτήσουμε καταλήλως. Όπως ε, είπε ο Βέρμαν, τα συστήματα bottom-up δεν ε, λειτουργούν επαρκώς στον τομέα της ανάπτυξης. Τα προγράμματα τα οποία ε, οργανώνονται top-down, όπου ε, τα οποία εκτελούνται από τις κυβερνήσεις δίχως να λαμβάνουν υπόψη τους μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους μη κρατικούς φορείς δεν αποδίδουν επαρκώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνένεση έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερο ε, διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο. Θα ήθελα να πω τώρα στην Κομισιόν. Πολλοί από τους παρόντες ε, την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της ε, Κοινοβουλικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ΑΚΕ, ο πρώην Επίτροπος Λουί αναγνώρισε ρητά πω ε, οι διαδικασίε και τα συστήματα διαχείρισης ε, της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ περίπλοκα, δυσκίνητα και δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από πλευρά αναπτυσσομένων χωρών και ειδικά από του μη κρατικού φορείς. Γι' αυτό λοιπόν παροτρύνω την Κομισιόν πως η αναθεώρηση της απλοποίησης που θα γίνει την επόμενη χρονιά να, ε, να τίνει προς ε, μεγαλύτερες αλλαγές, πιο βαθιές αλλαγές από πλευράς κομισιών έτσι ώστε να συνεχίσουν να εγγυώνται ότι δαπανούνται πόροι που, έχουν, που έχουμε για την ανάπτυξη αλλά να δαπανούνται πολύ πιο αποτελεσματικά διότι οι διαδικασίες είναι ε, ιδιαίτερα δύσκολες και δυσκίνητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Επέγκ από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, είμαι όμως αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής του Ελέγχου Προπολογισμού. Την ε, Παρασκευή είχαμε συζητήσει όλη την, ε, ε, όλη αυτή την προβληματική. Και θέλω να αναφέρω το ρητό που χρησιμοποιείται συχνά στην Ολλανδική λογοτεχνία, ότι από τα λόγια στα έργα απέχουμε παρασάγκας. «915 εκατομμύρια είχαμε το 2007, μια σημαντική αύξηση ε, των 100 εκατομμυρίων από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα στην απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Εγώ ως δημοσιογράφος επισκέφτηκα πολλές αφρικανικές χώρες και πρέπει να διαπιστώσουμε από κοινού ότι έχουμε φτάσει στα όρια της εφικτότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. Δεν μπορούμε εμείς να, λύσουμε όλα τα προβλήματα της, ε, της Αφρικής. Ε, θα έπρεπε σε για, για πολλά θέματα για πολλά ζητήματα να, να, να αναστείλουμε τις πληρωμές. Λένε 15.000 μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μα πού στο καλό είναι αυτές οι 15.000 μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πρόκειται δηλαδή για έναν τεράστιο τομέα ε, απασχόλησης ε, ε, προσωπικού. Έχουμε εμεί πίνακε γραφειοκρατικού χαρακτήρα με λεπτομέρειες και κόντρα λεπτομέρειες και λογιστικά στοιχεία κτλ. Και έχουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις από την άλλη μεριά που αντιμετωπίζουν όλες τις πρακτικές δυσκολίες. Και εντάξει να οργανώνουμε σεμινάρια και κατάρτιση. Αλλά πάντα θα έχουμε τα όρια που θέτει η λογική της συνεργασίας. Χαίρομαι λοιπόν που είμαστε διαθέσιμοι να εξετάσουμε το θέμα Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με λύσεις πιο διαρθρωτικές και όχι με απλουστευτικές λύσεις του τύπου περισσότερα λεφτά έχουμε τόσο το καλύτερο. Ο κύριος Ρισελ για να... Α, όχι, λάθος, λάθος. Έλεγα τρεις-τρεις ε, να, να μιλήσουνε. Ο κύριος Ρισελ, λοιπόν για να απαντήσει στις τρεις ερωτήσεις που ετέθησαν και μετά ξανά άλλος γύρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Έπινγκ είναι δύσκολο να πάρω πολιτική θέση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χρημάτων γιατί και εμείς βέβαια εμείς περιμένουμε να δούμε την απορρόφηση, πώς θα, θα δαπανηθούν. Γιατί σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο κύριος ε, Μπέρτμαν μου φαίνεται ότι ε, σοκαρίστηκε λίγο γιατί δεν ε, δώσαμε σαφείς και πλήρης ενδείξεις σχετικά με το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Και στις αντιδράσεις μας στην έκθεση του Ελεκτικού Συνειδρίου και στις συζητήσεις μας με τους υπεύθυνους από την ΕΚΟΚΟΜΠΗ ήδη έχουμε καταδείξει ορισμένα θέματα είναι ευρείε πολιτικές ε, μέχρι διαδικαστικά, από ευρείε πολιτικές μέχρι διαδικαστικά πράγματα. Για το τετραμερή διάλογο, αυτό το αναγνωρίσαμε, δεν ήταν όλοι στο Παλέρμο, αλλά είναι μια συζήτηση που, όπου συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών και τα κοινοτικά όργανα και οι κυβερνήσεις, αυτοί οι τέσσερις. Και θα πρέπει και μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών από τι νότιε χώρε θα πρέπει να συμμετέχουν. Γιατί αυτό δεν είχε γίνει τόσο πολύ την προηγούμενη φορά. Και βλέπουμε ότι και από τι θεματικέ γραμμέ του προπολογισμού το 70% που δαπανούνται είναι σε βόρειε μη κυβερνητικέ οργανώσει και όχι νότιε. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε. Γι' αυτό θέλουμε να συζητήσουμε, να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Να συζητήσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι θα βγάλουμε θα κάνουμε μια πρόσθετη προσπάθεια στον τομέα της δημιουργίας ικανοτήτων, γιατί υπάρχει η ζήτηση για αυτό το πράγμα. Όμως μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων πόρων που υπάρχουν, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε προσπάθειες μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να οριστεί αυτό ως αναπτυξιακή ε, δραστηριότητα καθ' αυτή και θα πρέπει να ε, βρούμε χρήματα για την εκπαίδευση κλπ. Και θα πρέπει να τα σταθμίσουμε, να δούμε θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα ή προτιμάμε να δαπανίσουμε ε, στους ανθρώπους στις στοχότερες χώρες τα χρήματα αυτά ή στην εκπαίδευση για αυτά τα θέματα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση υπέρ του Α ή Β να το κάνουμε. Αλλά υπάρχουν όρια. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και οι αντιπροσωπείες δεν είναι στελεχωμένες για να κάνουν τα πάντα. Για τις προτάσεις για την απλοποίηση. Πολύ καλά είπε ο κύριο Γκερέρο για τι διαδικασίε και για την Κομισιόν που πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει τι διαδικασίε προ το καλύτερο. Δεν θέλω να παίζουμε κρυφτούλι τώρα εδώ σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε τελευταία ανάλυση οι προσπάθειές μας καθορίζονται και σφραγίζονται από τη Δημοσιονομική Αρχή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο. Και την περασμένη φορά που μιλήσαμε για την απλοποίηση, σαν εν τη γενέση τους πολλές απλουστευτικές προτάσεις. Γιατί δεν υπήρχε η πρόθεση να γίνει αποδεκτή που και πολλή δημιουργικότητα από την Κομισιόν. Και αυτό και για τη λογοδοσία ισχύει. Και είναι και πολιτικό το θέμα επίσης εδώ. κυρία Πλάτη είπε πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στη λογοδοσία των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενε χώρε. Αυτά είναι δύο, διαφορετικά πράγματα. Πρέπει κανεί να λογοδοτεί για αυτά που κάνει και να σέβεται όμως την ιδιοκτησία των ανθρώπων σε μια πτωχή χώρα. Πέραν αυτού θα πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία για τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και αυτή είναι μια δουλειά η οποία θα πρέπει να γίνεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της αρχής επί του προϋπολογισμού. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε το ένα και να μην κάνουμε το άλλο και οι δύο λογοδοσίες πρέπει να υπάρχουν. Τώρα για την απλοποίηση δεν ε, πέρασαν προτάσεις πολλές, αλλά αν θέλουμε να ε, μιλήσουμε για ίσους κανόνες του παιχνιδιού, διαφάνεια κτλ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αλλάξουμε το σύστημα, ας πούμε, για την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Αν τους καλέσει κανείς όλους και τους δώσει ευκαιρία όλους, οι δημόσιες αυτές ε, συμβάσεις, οι κρατικές συμβάσεις είναι ανοιχτέ διαδικασίες, είναι καλύτερε. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και πολλή επαγγελματική ζήλια ε, εδώ. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν να μας σύρουν στα δικαστήρια διότι ε, δεν έγινε σωστά η διαδικασία, η αξιολόγηση κλπ. Και πολλές φορές ε, είναι επαχθής η διαδικασία γιατί μέσα από τις λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει κάθε φορά να δικαιολογούμε τη στάση μας γιατί κάναμε το α, το β κλπ. Νομίζω ότι απάντησα και στον κύριο Μπέρμαν και στον κύριο Γκερέρο και δεν απαντώ στον κύριο Έπιν γιατί είναι καθαρά πολιτικό το θέμα που έθεσε. Δεν είναι δικής μου αρμοδιότητας. Ο κύριος Βένσον έχει το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, επεξεργαστούμε όλη αυτή τη δουλειά, να την αναθεωρήσουμε σε μόνιμη βάση, γιατί όλα αυτά τα ε, δεδομένα είναι περίπλοκα και σύνθετα και δεν μπορεί να περιοριζόμαστε στην έκφραση μόνο επιθυμιών. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε την διαφάνεια, η οποία θα πρέπει σαν κόκκινη κλωστή να διατρέχει όλες τις δραστηριότητες των δωρητών, αλλά να υπάρχει και από τη μεριά των αποδεκτών. Ε, αυτή τη συζήτηση την ξέρω πολύ καλά και μέσα από το σουηδικό πρίσμα. Ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Σουηδία και ασχολήθηκα επί χρόνια για αυτό το θέμα. Και πολλές φορές οι μη κρατικές οργανώσεις ε, κάνουν δουλειά με πολύ πιο ορατό τρόπο από ό,τι κάνει ας πούμε η κρατική βοήθεια. Αυτό δεν πρέπει να μας αγχώνει, μπορεί να έχει και τις θετικές του πλευρές. Επίσης αναφέρθηκε εδώ ότι οι σχέσεις πρέπει να εμβαθυνθούν και ότι οι δύο εταίροι, εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, ούτω ώστε οι δωρητές και οι αποδέκτες να ε, αναπτύξουν μεταξύ τους ισχυρότερους δεσμούς να ε, αναβαθμίσουν και οι δύο τη θέση τους. Όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το ενδεχόμενο της ήτας. Ε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντοτε. Εκείνο που είναι σημαντικό πάντως είναι κάποια στιγμή να βγαίνουν προς τα έξω και επιτυχημένα προγράμματα. Και οι δωρητές που πολλές φορές, δεν, ε, που πολλές φορές κατακρίνονται θα μπορούν έτσι να δείξουν ότι βελτιώνεται διαχρονικά η συνεργασία και την ποιότητα των προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τα, τους εκπροσώπους των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Η έκθεση ήταν ενδιαφέρουσα αλλά ταυτόχρονα πολύ θεωρητική. Θα ήθελα να έχουμε μια μεγαλύτερη πρακτική χρειά σε αυτή την έκθεση. Η τεχνικότητα της έκθεσης δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε και την όλη πολιτική του διαβήματος. οι διάφοροι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να υπόκεινται τον έλεγχο της Κομισιόν ή των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει ήδη να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν την, ε, τις πρωτοβουλίες τους. Και από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Ρισελ, η Κομισιόν έχει τεράστιες δυσκολίες στο να θέσει υπό έλεγχο αυτούς ε, τους ε, μη κρατικούς ε, χρήστε. και αυτοί μπορούν να παίξουν έναν ουσιαστικότατο ρόλο στην ε, οικοδόμηση των ε, κοινωνιών στις υπανάπτυξη χώρες, κυρίως εκεί όπου δεν υπάρχει καμία κυβερνησία, όπου δεν υπάρχει οργανωμένη κρατική υπόσταση. Οι μη λοιπόν κρατικοί οργανισμοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιοχές, διότι αν φυσικά είχαμε μία οποιαδήποτε διακυβέρνηση σε αυτές τις χώρες, ε, ε, δεν θα χρειαζόμασταν και αυτού του είδους ε, τους οργανισμούς. Θα πρέπει να παίξουν λοιπόν ένα γεφυροποιό ρόλο εκεί όπου δεν υπάρχει κρατική οργάνωση και δημοκρατία. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ε, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, μην το ξεχνάμε, παίζουν έναν τεράστιο ρόλο ε, ε, χρηματοπιστωτικής πλαισίωσης. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι πάρα πολλά λεφτά και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό συνολικά για ε, τις ανάγκες ε, της αναπτυξιακής προσπάθειας. Εγώ θα ήθελα να ξέρω όμως τι λένε και τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία ελέγχουν και τα ουσιαστικά ε, σημεία της αναπτυξιακής πολιτικής. Η Κομισιόν σε όλα αυτά παίζει έναν συντονιστικό ρόλο. Δεν μπορούμε εμείς ε, να είμαστε υπόλογοι για τους μη κρατικού οργανισμούς, άμα αυτοί δεν χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αλλά δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι χρηματοδοτούνται και από τα κράτη-μέλη. Για τους ελέγχους τώρα, ο πολύς έλεγχος είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός, αλλά χωρίς ε, έλεγχο ε, διατρέχουμε τον ε, κίνδυνο ε, να, να, έχουμε απώλειες. Δηλαδή, ο, ο πολύς έλεγχος εν τη γεννήση του καταστρέφει ένα σχέδιο. Διότι όντας μικρές ε, διαρθρώσεις αυτές που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του σχεδίου με τον πολύ έλεγχο δεν μπορούν να συνεχίσουν. Τώρα, το να μην έχουμε αρκετό έλεγχο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και εδώ να αναφέρω κάτι το πάρα πολύ πρακτικό. Εγώ είχα ε, στον, ε, στον καιρό μου, υπό την ευθύνη μου, ε, ντοσιέ για αυτά τα θέματα. Και υπήρχαν 100.000 έλεγχοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ε, από τα κράτη δικαιούχους κλπ και στο τέλος διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι τι είχαμε ανακαλύψει, ανακαλύψει ότι υπήρχε δυνατότητα διπλής χρηματοδότησης, δηλαδή ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί για χρηματοδότηση στην Κομισιόν και ταυτόχρονα είχε κατατεθεί και στο, στο Εθνικό Κράτος. Υπήρχε λοιπόν αυτή η διπλή κατάθεση του σχεδίου και εδώ μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα. Τώρα, ένα άλλο σημείο για να είναι πιο πρακτική η συζήτησή μας θα ήθελα να υποβάλω την εξής πρόταση. Μήπως μπορούμε να βασιστούμε σε έναν κύκλο σχεδίων. Λοιπόν, το σχέδιο πότε ξεκινάει. Όταν ε, στο μυαλό ενός ε, ε, εθνικού εταίρου του μπαίνει η ιδέα να συνεργαστεί με μία νότια χώρα. Αν λοιπόν αυτή η σπίφα ε, προκύψει το 2009, τότε η υλοποίηση του σχεδίου τελειώνει το 2020. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς από τα σχέδια του 2009 να τα δούμε κυκλικά, για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η αχίλιος πτέρνα όλης αυτής της διαδικασίας. Και επειδή πολλοί από εμά είναι νέοι βουλευτές, και εγώ είμαι καινούριο σε αυτήν την Επιτροπή, Πώς, να πώς λοιπόν οι μη κρατικοί φορείς θα μπορούν να εργάζονται υποκείμενοι στους απαραίτητους ελέγχους, οι οποίοι όμως δεν θα πρέπει εν τη γεννήση της να καταστρέφουν την πρωτοβουλία και την υποβολή του σχεδίου. Επίσης, οι κρατικοί φορείς δεν θα πρέπει να επιβάλλουν στους μη κρατικούς φορείς και στους μη εθνικούς φορείς μεθόδους που δεν στέκουν. Χρειάζονται μέθοδοι που να είναι αποτελεσματικές, γρήγορες και αηφόρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο σημείο που είχα να πω. Τώρα, να ρωτήσω την Κομισιόν. Όταν υπάρχει πρόβλημα, όταν υπάρχει διαφωνία με τους εταίρους, μεταξύ των εταίρων, και έχετε κράτη-μέλη από τη μια και χώρες και από την άλλη. Τι κάνετε, αντιμετωπίζετε προβλήματα αυτού του τύπου, δηλαδή όταν έχετε μία χώρα δικαιούχο η οποία δεν θέλει τον μη εθνικό φορέα που εργάζεται στην επικράτειά της. Πώς τη λύνεται αυτή τη διαφωνία. Και κάτι άλλο, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Έχετε ανθρωπιστική βοήθεια ε, με στόλους και ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς στολή. Αν είχατε εσείς στο Αφγανιστάν μη ενστόλους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και έχετε και τους στρατιωτικούς ε, δεν πιστεύετε ότι πολλές φορές η πολιτική, η μη ένστολη τέλος πάντων της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν τα αντίπεινα και την ύφη για τη στρατιωτική παρουσία. Πρέπει να λύσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και να πούμε στους διάφορους εθνικούς ε, φορείς ότι μην υποσκάπτεται την ε, παρουσία των ανθρωπιστικών οργανώσεων στις χώρες αυτές. Διότι η στρατιωτική παρουσία κάποια η ανθρωπιστική βοήθεια όμως συνεχίζει να υπάρχει ως ανάγκη και οι ανθρωπιστικές, ελπίζω και αυτή κάποτε να σταματήσει βεβαίως να υπάρχει ως ανάγκη, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις μέχρι να τελειώνει αυτή η ιστορία πρέπει να είναι εκεί και να παλεύουν. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο σε μένα την ίδια για να ρωτήσω και εγώ κάτι την Κομισιόν. Η διαδικασία του Παλέρμου, η διαδικασία διαλόγου μεταξύ Κομισιόν, Κοινωνίας των Πολιτών και του Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχει μια νέα όθηση μέχρι το 2010. Λοιπόν, ρωτώ την Κομισιόν, τι μέτρα έχετε λάβει ώστε αυτός ο διάλογος να καρποφορήσει. Και τώρα να δώσω το λόγο σε άλλους δύο εμπειρογνώμονες που δεν μίλησαν και μετά η Κομισιόν απαντήσει συνολικά στις ερωτήσεις. Ο κύριος Κίνστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αν κατάλαβα καλά, έγινε και απευθείας ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Τονίζω λοιπόν ότι ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας που ξέφρασαν εκτίμηση για το έργο μας. Δεν θέλαμε να σοκάρουμε κανένα με το περιεχόμενο του ελέγχου και ελπίζω να μην σας δώσαμε μια θεωρητική και μόνο έκθεση ε, ελπίζω να μπορέσαμε να κρίνουμε θετικά αυτά που ήταν θετικά σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της Κομισιόν για τη συνεργασία και όμως από την άλλη κάποιες αδυναμίες και κενά. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν η έκθεση βοήθησε να αρχίσουν κάποιες βελτιωτικές διαδικασίες και δεν ήταν κάτι εντελώς ε, ε, καινούριο χωρίς δηλαδή αναφορά στην πρακτική εφαρμογή. Για την απλούστευση της διαδικασίας ε, δεν θεωρούμε ότι μια απλούστευση ε, ντε και καλά είναι πάντα υπέρ της διαφάνειας ή της νομιμότητας των συνεργασιών. Επίσης, ε, δεν θέλω να επισέλθω στις ερωτήσεις των συναδέλφων σχετικά με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Υπάρχει, ε, ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες χρηματοδότησης και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικές εκεί όπου οι μη κρατικοί φορείς θεωρούνται εταίροι και θεωρούνται και οι, η αρχή ή που υλοποιεί το πρόγραμμα. Εμείς ε, οι ελεγκτές ε, θέλουμε ε, πάντοτε να ελέγχουμε τις διαδικασίες μετά. Δηλαδή, όπως λέμε, θέλουμε να μετράμε τα, τους λαγούς μετά το κυνήγι. Δύο-τρία χρόνια μετά κάνουμε ένα follow-up ή μάλλον κρίνουμε ποιο follow-up, τι συνέχεια έδωσε η Κομισιόν στις παρατηρήσεις μας. Και αυτό μάλιστα προτιθέμεθα να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση για να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πλάτ. Πολλά θέματα θα ήθελα να σχολιάσω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και θα παρουσιάσω κάποιες προσωπικές απόψεις. Χαίρομαι πολύ που τόσοι πολλοί άνθρωποι και ο κύριος Γκερέρο μας υπενθύμησαν ότι αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι πολύ σημαντική αναπτυξιακή δρόντες ή μη κρατικοί φορείς. Εγώ δεν το νιώθω αυτό ως μη κρατικός φορέας, δηλαδή δεν το αισθάνομαι, δεν με κάνουν να το νιώσω ότι με θεωρούν σημαντική στο, στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές διαιρωτώ με αν είναι τόσο σημαντικό αυτό, γιατί είναι τόσο δύσκολο να, ενταχθούν οργανώσεις της κοινωνίας των, πολιτών, των ε, και από τον Νότο στην προγραμματική διαδικασία. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τις ε, ε, διαβουλεύσεις, ώστε να προετοιμάζονται όλοι επαρκώς πολλές φορές ε, ακούμε αρνητικά πράγματα για την παρουσία των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις, ενώ πολλές φορές δεν τους δόθηκε ο χρόνος για να προετοιμαστούν καλά. Και αυτό παίζει ρόλο σε σχέση με την ε, δημιουργία ικανοτήτων. Ε, ακούσαμε κάποιες συστάσεις σε σχέση με το βασικό προσωπικό και τις αντιπροσωπίες και συμφωνούμε ότι χρειάζεται, χρειάζεται μόνιμο προσωπικό που θα μπορεί να δουλεύει και να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ένας οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που είναι σύνθετο πράγμα και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επίσης, ε, ποιες, οι πιο αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις ε, σημειώθηκαν σε περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να συνεργαστεί στενά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σημειώνω επίσης ε, μια δήλωση που έγινε στην αρχή ότι όταν δούμε τα χαρακτηριστικά των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά στον προβληματισμό μας, στον προβληματισμό μας στο μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή να παίζει ρόλο πολύ σοβαρό ε, η κάθε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση. Είμαι βεβαία ότι χάνομαι, διασπαθίζομαι ε, και τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη και ανθρώπινους πόρους από την κοινωνία των πολιτών γιατί δεν ξέρουμε να τις ε, αξιοποιήσουμε, να τους αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Κύριε Ρουσέλ, δεν άκουσα. Τι είπατε αυτό το 70% του χρηματοδότηση που πάει σε βόρειες, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, το 50% ε, εάν πήγαινε στις οργανώσεις αυτές, στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, θα είχαμε ε, μια καλύτερη ισορροπία. Μου φαίνεται ότι πρέπει να τροποποιήσετε λίγο τις στατιστικές σας. Ε, επίσης, ε, άκουσα γι' αυτό που, και χαίρομαι ε, που είπατε ότι στηρίζομαι την καινοτομία στους μη κρατικούς φορείς, κοινωνία των πολιτών προσπαθούμε εμείς. Εμείς πολλές φορές παίζουμε πολύ ενεργό ρόλο, αλλά και σε σταθερές χώρες, όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες καινούργιες χώρες, μπορούμε και στην περίπτωση όπου υπάρχει σταθερότητα, να συνεργαστούμε με τις ε, ε, σταθερές κυβερνήσεις και να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικά προγράμματα. Επίσης, ε, δεν υπάρχει ρίσκο στη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα λογοδοσίας, αλλά αυτό είναι κάτι που το παρακολουθούμε πολύ σε όλες τις δράσεις, είτε χρηματοδοτούνται από ιδιώτες δωρητές ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας είναι πολύ σημαντικό θέμα και την ευθύνη μας εδώ την παρακολουθούμε, θέλουμε να βελτιωνόμαστε, είμαστε ε, ένα, αν θέλετε, ε, ετερόνυμο πλήθος οργανώσεων η μία καλύτερη, η άλλη χειρότερη, δεν έχουμε όλοι το ίδιο επίπεδο και άρα μας ενδιαφέρει αυτό. Τώρα, για την ιδρώντες στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών δεν έχουν κανένα πρόβλημα να απορροφήσουν μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης αν θελήσει να αυξήσει τη βοήθεια η Επιτροπή. Ο κύριος Ρισελ για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. έγιναν πολλές παρατηρήσεις ε, ποικίλη φύση. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναρθούμε με ποιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούμε να συζητάμε και να διαπραγματευόμαστε. Εμείς τους έχουν γίνει επιλογές, γνωρίζω κράτη και τα οποία έχουν αποφασίσει να συνεργάζονται με έναν μικρό αριθμό μη, κρατικών φορέων. Αυτό εντάξει δεν είναι ένα πρότυπο το οποίο επιλέγει όμως για την Ευρώπη. Εμείς ε, θα πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε διαδικασίες ε, πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με όλους ε, για να παρέσει τον κύριο Γκόλτ, ε, ναι, όντω με κατανόησε σωστά ότι δηλαδή μη κρατικοί φορείς δεν θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη σκέπη της Κομισιόν. Εμείς υποβάλλουμε πρόσκληση υποβολής πρότασης ε, και όποιος έχει λαμπρές ιδέες ε, για οποιαδήποτε χώρα οι ιδέες αυτές είναι πρόσδεκτες. Όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη μέθοδος, δηλαδή να λάβουμε υπόψη ότι φέτα, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των παιδιών στις ε, τενεκιδοπόλεις. Λοιπόν, ε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν περιρίζεται τον ε, αριθμό των προγραμμάτων είναι φυσικά πολύ πιο εύκολο να συγκριθούν κλπ. Αλλά δεν επιλέγεται κάτι τέτοιο. Εμείς ε, κάνουμε μια διαδικασία ανοιχτή σε πρόσκληση υποβολή προτάσεων, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και μετά φυσικά δεν μπορούμε όλες να τις ε, χρηματοδοτήσουμε διότι πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Ε, είναι θέμα επιλογής λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αυτή την ανοιχτή διαδικασία, ε, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ε, πολλοί ένδυνα υποψήφοι και σε ό,τι φορά την αποτελεσματικότητα έχουμε κάποια προβλήματα ομολογουμένως. Ο κ. Γκέρνς ε, μίλησε για το τι κάνει η Κομισιόν και τι κάνει η Μέλη. Ειλικρινά δεν γνωρίζω διότι αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ε, των Βρυξελών, δηλαδή τι κάνει η Κομισιόν και τι προγραμματίζει να κάνει. Δεν υπάρχει φόρουμ στην ε, Βρυξέλλες όπω συζητάμε για ένα κράτο. και όταν συζητάμε για προγραμματισμό και αυτό λέω προ την κυρία Πλάτ οι μη κυβερνητικοί φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα προγραμματισμό ο οποίος ε, έχει σχέση με αυτόν της Κομισιόν και δεν υπάρχει κάποιο φόρουμ για να μπορέσει να ζητηθεί Αυτό είναι ένα από τα δύναμα σημεία του όλου συστήματος. Με λίγα λόγια λοιπόν, κάποιος θα μπορούσε να πει από τις μη κρατικούς φορείς ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ασχοληθεί με τα ζητήματα υγείας και το τι κάνουν οι υπόλοιποι φορείς εκεί. Νομίζω λοιπόν πως ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει κατάλληλο συντονισμό των δωρητών και να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του προγραμματισμού και να υπάρξει συμμετοχή των ε, κοινωνία των πολιτών σε αυτή την ολιστική προσέγγιση. Αυτά βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με τα όσα ανέφερα για την ατζέντα της Άκρα και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αλλά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ούτε στις Βρυξέλλες σε θέματα συντονισμού προγραμμάτων. Ο κύριος Γκιόνης επίσης αναφέρθηκε στον έλεγχο, ότι υπερβολικός έλεγχος ε, ε, δεν ε, είναι αποτελεσματικός και ο λιγοστός επίσης. Χρειάζεται λοιπόν να χειρίσουμε κάποιες Κάποιε αποστάσει. Ε, το επίπεδο του κινδύνου θα πρέπει να υπολογίζεται και στην ουσία θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνο ε, στα όσα κάνουμε. αλλά ξέρετε πως ε, η ανάπτυξη ενέχει και, του, και κινδύνους. Αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά χρονικά όρια και περιορισμούς, ναι, πρέπει να δεσμεύσουμε τα χρήματα στην περίοδο νήσιν 1. Λοιπόν, αυτά τα οποία θα πάρουμε για το Δεκέμβριο 2010 θα πρέπει να δεσμευτούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα το τέλος του 2010. Διαφορετικά θα απολαστούν και όταν δεσμευτούν μέσα σε αυτό το νήσιν 1 χρονικό όριο, τότε μέσα σε τρία χρόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά το πρόγραμμα καταραίει. Με αυτό αναφέρεται στους κανονισμούς και ειλικρινά αυτό θα πρέπει να το τηρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από την φιλανθρωπία. Η ανάπτυξη σημαίνει και business. Αν υπάρχουν λοιπόν προγράμματα θα, τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα σε συγκεκριμένα προθεσμίες και περιθώρια έχει αλλάξει κάπως η μορφή και η κουλτούρα της ε, ανάπτυξης, αλλά τι να κάνουμε. Μπεστούση πρέπει να φροντίσουμε να μην κάνουμε σφάλματα και να βρισκόμαστε πάντα από, μια, από κάποια πίεση προκειμένου να ε, ολοκληρωθεί το έργο ή το πρόγραμμα. Τώρα, παρατηρήσει σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια με ένστολους ή χωρίς Ξέρετε πως ε, υπάρχει το, η δήλωση η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να δίνεται με ε, δεν να χορηγείται από ένστολους αλλά εδώ και χρόνια έχει αλλάξει η νοοτροπία και έχουμε τα 3D ε, Development, Democracy and Defense διπλώματος συγγνώμη και όχι δημοκρασία ε, προσωπική μου άποψη είναι πως ε, θα πρέπει να έχουμε, αποκτήσουμε την οτροπία της σύγχρονης ε, ανταξιακής βοήθειας Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι το πεδίο εδώ είναι επικίνδυνο και ολιστήρο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια καθαρή ιδέα σχετικά με το που θέλουμε να πάμε τώρα. Σε ό,τι αφορά το Παλέρμο, θα οργανώσουμε έναν τετραμερή διάλογο του 2010 και είναι σαφέ πω η ατζέντα θα πρέπει να είναι ευρύτερη δυνατή. Το τι θα σημαίνει το Παλέρμο, αυτό εξαρτάται και από του συμμετέχοντε. Αν θέλουν να συζητούν κανένα ζήτημα, τότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μία συνεδρίαση και παφ, τελειώσαμε. Ε, πρέπει λοιπόν να, να ζωγονίσουμε αυτόν τον ε, τετραμερή διάλογο, διότι βρισκόμαστε στο πλαίσιο της ενδιάμεση αναθεώρησης. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και αυτά τα θέματα και καταρχήν η ατζέντα θα πρέπει να αφορά στο μέλλον θα πρέπει να οργανώσουμε τι θα συμβεί μετά το 2013. Συνήθω αυτό ο προγραμματισμό ξεκινάει δύο χρόνια νωρίτερα. 2010-2011 λοιπόν είναι χρονιέ πάρα πολύ σημαντικέ για τον διάλογο αυτό. Αλλά αυτά τα οποία βρίσκονται στην θα βρεθούν στην ατζέντα εξαρτάται και από του υπόλοιπου εταίρου μα στο πλαίσιο του διαλόγου. Τώρα, το θέμα του σημείου επαφή για κάθε προσωπία για κάθε μη κυβερνητική οργάνωση, θα να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλο για κάθε ε, μη κρατικό φορέα και τις σχέσεις μας, αλλά ευαισθούς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα για τις στατιστικές, 70% του θεματικού προπολογισμού είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε από διαδικασία διαδικασίες πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Εάν δεν και όλα αυτά καταδεικνύουν ότι κυβερνητικές ε, ευρωπαϊκές, ε, κρατικοί ευρωπαϊκοί φορείς λαμβάνουν μέρος ε, και Μπορώ κάλλιστα να θέλει, να σας δώσω πληροφορίε αναφορικά με αυτές τις ε, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων οποιαδήποτε στιγμή δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητήσατε το λόγο. Λοιπόν, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση μεταξύ του κυρίου Ρισελ ε, και μου, να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Εγώ εδώ ε, εξέφρασα μία πεποίθηση. Είπα ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η αυτονομία δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλοι έχουν ένα ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα που εκφράζεται στη συζήτηση. Πρέπει να αναπτύξουμε μία κουλτούρα του ρίσκου. Αν εμείς εδώ θεωρήσουμε ότι πρέπει να αναπτύσσουμε πολιτικές χωρίς να ρηψοκινδυνεύουμε τίποτα, τότε γινόμαστε όλο ένα και λιγότερο πιο ευρηματικοί. Και οι κανόνες θα, θα, θα, είναι στήρι κανόνες εφαρμογής δημοσιονομικού ελέγχου. Ο πολλής έλεγχος σκοτώνει τη φαντασία, την πρωτοβουλία. Πρέπει λοιπόν εμείς να προωθήσουμε αυτήν την κουλτούρα του κινδύνου και να την καλλιεργήσουμε. Διότι το αν, αν αναλαμβάνουμε εμείς πολιτικές με μηδενικό κίνδυνο, αυτό δεν έχει κανένα όφελος για το μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους μας ε, ε, του Νότου διότι ξέρουμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε στις χώρες μας δεν μπορούν να εφαρμόζονται ε, ακριβώς ίδιες στις χώρες του Νότου. Εμείς ε, εργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, με τη λογική της διαφάνειας κλπ. Τώρα, πού μπορούν και πώς μπορούν να πλαισιωθούν οι μη κυβερνητικές και οι μη εθνικές οργανώσεις. Πού μπορούν να ταξινομηθούν, σε, σε ποια κατηγορία. Θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται και είναι και το πιο λογικό εδώ στις Βρυξέλλες ή στις χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για την στρατηγική κατά τη φτώχεια σε εθνικό επίπεδο εμείς ε, καλούμε οργανισμούς ε, του ΟΗΕ Σε αυτά τα φόρουμ λοιπόν υπάρχει θέση για τους μη εθνικούς φορείς. Αν δεν έχει προβλεφθεί, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε μία θέση και για αυτές τις οργανώσεις και να καταλάβουν αυτή την κατάσταση και να βρούνε όμως και τη θέση τους μέσα σε όλη αυτή τη διάταξη μέτρων. Ευχαριστώ για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είναι στη φύση των ε, εκθέσεων του ελεκτικού συνεδρίου να είναι προκλητικές. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας όμως όλα αυτά τα στοιχεία και παρακαλούμε την ομάδα εργασίας D, Δέλτα, για, τους, ε, για την κοινωνία των πολιτών να αναφέρουν σχετικά διότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι το 1% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί έχω τις σημειώσεις μου στα αγγλικά. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, τροποποίηση του μέσου σταθερότητας. Έχω μια πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού 17-2006 που θεσπίζει ένα μέσο σταθερότητας εισηγητής ως εισηγητής μάλλον σκέφτηκα να ασχοληθώ με δύο ζητήματα. Αφενός το θέμα των ε, φορητών όπλων, τον κανονισμό, εξού και η απόφαση που από την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αφετέρου, έχω προτείνει μια τροποποίηση σχετικά με το ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δυναματίζει στον τομέα τη οικοδόμηση ειρήνη και την επίλυση των σειράξεων. Ε, αναφέρεται ανώτατο όριο 5% πόρων που παρέχονται για την καταπολέμηση της διάδοσης φορητών όπλων και φορητού εξοπλισμού Προτείνω επίσης ε, για μια οικοδόμηση μέτρων ε, μέχρι με 5-10%. Θα δώσω να δώσω τώρα το λόγο λοιπόν στα μέλη που θέλουν να σχολιάσουν το ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε βασικά θα ήθελα να υποστηρίξω το νόημα αυτής της τροπολογίας που έχει κατατεθεί. Εγώ ως ε, καθηγητής ε, πολιτικών επιστημών αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στα θεσμικά όργανα από ότι στα άτομα και στην ε, τακτική λειτουργία των κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και στην πολιτική κουλτούρα από ότι στα ατομικά συμφέροντα. Και θεωρώ λοιπόν πως ε, εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες που έχουν αδύναμους θεσμούς να τους υποστηρίξουμε λοιπόν, διότι θεωρώ πως πρόκειται για μια δομή που βοηθάει στην ανάπτυξη αυτών των κοινωνιών, αλλά και καθενός από τους πολίτες τους, διότι οι θεσμοί είναι αυτοί που μεταδίδουν τις λειτουργίες της δημοκρατικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου λοιπόν υποστηρίζω αυτή την τροπολογία για τον ανώτατο όριο του 10%. Ούτε σε έχει ζητήσει το λόγο, κλείνει το μικρόφωνο της Προέδρου. Δώσω το λόγο στον κύριο Καρκούιτε από τη Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρουσίαση θα κάνω των στοιχείων της τροπολογίας που είναι κομμάτι, ίσως ξέρετε, της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού μέσου ρέλεξε, εξωτερικών υποθέσεων. Ε, τον Απρίλιο έχει γίνει μια ανακοίνωση της Κομισιόν, την, την παρουσίασε στην προηγούμενη Επιτροπή η κυρία Φερέρο Βάλτνερ και συνοδεύεται από τρει νομοθετικού περιεχομένου προτάσεις για, που τροποποιούν τα υφιστάμενα κείμενα των νομοθετημάτων για το ICI, το DCI και το IFS με εξηγήσει από κοντά γιατί θεωρεί ότι χρειάζεται η Κομισιόν όλο αυτό το πράγμα για να ε, βελτιωθεί η εφαρμογή των μέσων. Για το μέσο σταθερότητας, το ε, εξηγηματικό memorandum στον κανονισμό προβάλλει το σκεπτικό ότι οι πρώτες, ε, οι πρώτες ε, τροπολογίες αφορούν τις αρμοδιότητες της Κομισιόν στα πλαίσια των κοινοτικοποιημένων πολιτικών και το μέσο σταθερότητας προκειμένου να λαμβάνουν δράση κατά της εξάπλωσης μικρών όπλων και οπλισμού κλπ. Αυτό είχε αποφασίσει να μην το κάνει η Κομισιόν μέχρι να έρθει η σχετική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση ECOWAS, ίσως την ξέρετε. Ήταν περσινή απόφαση και μετά την απόφαση συμφωνήθηκε ότι θα έκανε κάποιες αναπροσαρμογές ε, προτάσεις, δηλαδή αναπροσαρμογών ή ε, κομισιόν στο άρθρο 3 του κανονισμού για την ε, κρίση και την ετοιμότητα αντιμετώπισης κρίσεων και το άρθρο 4 του μέσου. Θέλαμε λοιπόν να ε, προσθέσουμε τον ελαφρύ οπλισμό και τα ελαφρά όπλα που δεν υπήρχε στο κείμενο πριν και να ενισχύσουμε τον τύπο και πεδίο εφαρμογής και το εύρος δηλαδή της δράσης που θα μπορούσε να προβλεφθεί και στα πλαίσια του μέσου σταθερότητας. Μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το σημείο παράλληλα γίνονταν συζητήσεις στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και έγινε εντατική η συζήτηση και αντιπαράθεση εκεί, γιατί μπορείτε να φανταστείτε ότι όλα αυτά γίνονται στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Είναι στο προσκήνιο ε, της δράσης και χρειάζονται και άλλες ε, συζητήσεις στο Συμβούλιο για τις τροπολογίες αυτές. Αυτά επί του παρόντος μπορώ μόνο να πω. Οπωσδήποτε δεν θα αντιταχθούμε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα. Οι άλλες δύο τροπολογίες που προτείνουμε αναφέρονται στο γεγονός ότι πρώτον η χρηματοδότηση, το όριο χρηματοδότησης για δράσεις στα πλαίσια του 4.1, δηλαδή διαπεριφερειακές απειλές της ασφάλειας, που είναι ευρύτατος ορίζον δράσης και ένα μακρότατο άρθρο περιορίστηκε στο 7% όταν εγκρίθηκε το μέσον το 2006. Το 7% για να σας δώσω μια ιδέα, μεταφράζεται σε μέγιστον 140 εκατομμύρια ευρώ σε μια επταετία, δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δράση σε 8 ή 9 διαφορετικούς τομείς περιφερειακού και διαπεριφερειακού επίπεδου. Δηλαδή, ε, πράγματα που η Κομισιόν δεν μπόρεσε να τα ε, ολοκληρώσει λόγω των ε, περιορισμών του προϋπολογισμού, όπως για παράδειγμα απειλές στις διεθνείς μεταφορές, κρίσιμες μεταφορές, ε, μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, κατανομή ενέργειας, επιδημίες, ε, απειλές στη δημόσια υγεία, ε, προκατεπίγουσες καταστάσεις, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, συνεργασίες, πράγματα δηλαδή τρέχοντα ή ε, συνεργασία με του ιού αυτής της γρήπης των χείρων, βοήθεια αντιμετώπισης, ε, προετοιμασίας όταν δεν υπάρχουν στις χώρες τα μέσα που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Προτείνουμε λοιπόν να αποκτήσουμε πιο πολύ ευελιξία, να πάει το κατόφλιο στο 10% που θα μεταφράζεται σε πρόσθετα 40-50 εκατομμύρια που θα διατίθενται την επόμενη τετραετία, ούτω ώστε να υπάρξουν και να υλοποιηθούν σημαντικά προγράμματα και να μπορέσει η Κομισιόν να κάνει μια διαφορά στον τρόπο χειρισμού όλων αυτών των θεμάτων που αποτελούν ε, πιθανές απειλές διαπεριφερειακές. Η πρόταση επίσης ε, και κάποιοι άλλοι, άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις άλλων χωρών να, να συμμετέχουν σε δράσεις του 4-3, δηλαδή προετοιμασία, ετοιμότητα που τα βάλαμε σε μια ομπρέλα, είναι, ομπρέλα είναι η εταιρική σχέση για την οικοδόμηση της ειρήνης με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη για την ε, συνεργασία, επιμερισμό γνώσεων κλπ. για την αντιμετώπιση ικανοτήτων από την Ελβετία κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν συμμετείχαν στις προκηρύξεις ε, ε, γιατί δεν είναι ε, τυπικά μέλη του EEA και δεν μπορούν να συμμετέχουν ενώ υπάρχουν πολύ ωραίες οργανώσεις, άριστες δίκτυα πρόληψης κρίσεων, διευθέτησης κλπ με τις οποίες συνεργαζόμεθα σε άλλα φόρα Άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί ο περιορισμός που προβλέπεται στην ένταξη του μέλους για να βελτιωθεί η συνεργασία με αυτές. Και τέλος για να κλείσω υπάρχει και η πρόταση παράλληλα να... Η πρόταση για το αύξηση του μεριδίου από 5 σε 10% σε αυτό το άρθρο του, ποσού, του ποσοστού. Να σας πω πού βρισκόμαστε. Το 5% μέγιστο μερίδιο όταν είναι ας πούμε 2 δις 62 εκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια το ποσό μεταφράζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην 7 ετία για δράσεις στα πλαίσια αυτού του άρθρου. Ήδη ήταν 5%. Και μέχρι τώρα δεσμεύτηκαν τα πρώτα δύο χρόνια 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορροφηθούν και 80 εκατομμύρια στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν προτάσεις και να αναλυθούν ε, οι δεσμεύσεις υποχρεώσεων. Κατά μέσον όρο 20 εκατομμύρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, για τα προγράμματα αυτά. Ήταν αυτό θα ήταν μια καλή στρατηγική. Το 5% ήδη αποτελεί σημαντική πρόκληση και για μας και για τους εταίρους μας από την κοινωνία των πολιτών, ώστε η ειρηνευτική αυτή εταιρική σχέση να δώσει από καρπούς. Έχουμε δε καλέσει και θα καλέσουμε εταίρους που δραστηριοποιούνται στις ειρηνευτικές διαδικασίες και είναι στις Βρυξέλλες και αλλού για οι πρώτες διαβουλεύσεις 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες πρώτη συνάντηση για να συζητήσουμε προτάσεις για του χρόνου και του παραχρόνου και τα αποτελέσματα μιας ανασκόπησης αυτής της εταιρική σχέσης στα πλαίσια των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών. Είναι η προσέγγιση μας και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να προειδοποιήσουμε λιγάκι. Δηλαδή ακόμα και να ανεβάσουμε το κατόφλι και το πάμε στα 10% μπορεί να μην τα καταφέρουμε και ούτε να χρειαστεί να, να δαπανίσουμε ε, το 5% που για να εξαντληθεί θα πρέπει να δώσουμε τα επόμενα χρόνια συν 80 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κρίμα που δεν δεσμεύσαμε παρά 20 εκατομμύρια ευρώ σε, αυτό, αυτή τη θέση, δεδομένου των μεγάλου αριθμού σειράξεων ανά τον κόσμο και τι τεράστιε ανάγκε που υπάρχει προκειμένου να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και θεσμού περιφερειακού. Θεωρώ λοιπόν πω δεν θα δυσκολευτούμε στο να χρησιμοποιήσουμε με τρόπο ικανοποιητικό το 10%. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί των υπολείπων προτάσεων της Κομισιόν, να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ε, πως ε, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι έχετε προθεσμία για να κάνετε τις ε, προτάσεις των Alors, Nous allons continuer. Θα συνεχίσουμε με το σημείο 8 της Μεσίας Διατάξεως. Πρόκειται για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις ε, βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Ας ε, δούμε λοιπόν τώρα την πρώτη τροποποίηση του κανονισμού 1943-2006 που θεσπίζει ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις ε, βιομηχανικές χώρες ε, και με άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος. Δυστυχώς ο κύριος Ντέβα δεν μπορεί να παραστεί σήμερα στις Βρυξέλλες που είναι και συγγυρής για να μας κάνει την παρουσίαση λόγω του συνεδρίου του κόμματό του. Ήταν αδύνατο να βρούμε κάποιον από την πολιτική ομάδα του κ. Ντέβα προκειμένου να τον αντικαταστήσει. Αλλά δεν θα θέλαμε να μεταθέσουμε την συζήτηση, διότι η αρμόδια τη Επιτροπή ΙΝΤΑ ε, πρόκειται να εγκρίνει το, την έκθεση. Και ο κ. Ντέβα δεν ε, διαφώνησε στο να κάνω εγώ την παρουσίαση. Μου έχει υποβάλει ένα κείμενο το οποίο και θα αναγνώσω εξ ονοματός του. Ιδού λοιπόν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί απάντηση στο ερώτημα του Κοινοβουλίου και ειδικά της Επιτροπής Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει μέτρα σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, που ξεπερνούν τα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθεια. Θέλουμε να προωθήσουμε ε, ε πρωτοβουλίε, συγγνώμη, για την αναπτυξιακή κομισιόν υποσχέθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει τέτοιε δραστηριότητε με βάση αυτό το κανονισμό, διότι δεν υπάρχει ελληνική βάση. Η Κομισιόν είχε αντιρρήσεις και το Κοινοβούλιο τόνισε ότι τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται από το μηχανισμό αντιλήψης συνεργασία θα πρέπει να συμβάλλουν προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι στόχοι μεταξύ αυτών η εκρίζωση τη φτώχεια. Η πρόταση που συζητάμε σήμερα ε, γνωρίζει αυτό το κενό που υπάρχει, αυτό το χάσμα που υπάρχει. Η Κομισιόν θέλει να δημιουργηθεί μια νέα νομική βάση προκειμένου να μπορέσουν οι οι αναπτυσμένες χώρες να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες και να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς να υπάρχει καμία στρέβλωση στο DCI. Το σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Ντέβα καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν και προτείνει μόνο μία τροπολογία. Αυτή η τροπολογία αφορά την χρηματοδότηση των ε, μη αναπτυξιακών μέτρων με, τον, ναι, νέα νομική βάση. Η Κομισιόν προτίθεται να χρησιμοποιήσει 180 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προβλέπονται για το μέσο του DCI. Η Κομισιόν τονίζει ότι ε, τα κονδύλια τα οποία χορηγούνται μέσω του προπολισμού στο DCI, δηλαδή 17 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013, δεν πρόκειται να μειωθούν αλλά η Κομισιόν θα προτείνει περαιτέρω πόρους ε, επιπρόσθετους από, για τους στόχους ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική και την Ασία. Και την περίοδο 2007-2013 η Κομισιόν έχει ανακοινώσει μία μείωση της τάξης των 100 εκατομμύριων ευρώ για το DCI. Το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κ. Ντέβα έχει αντιρρήσεις ε, σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό των κονδυλίων. Κάθε κονδύλι είναι απαραίτητο και θα πρέπει να ε, δοθεί σε άλλους, ε, σε άλλα τμήματα πέραν της ανάπτυξης. Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει κίνδυνος, ε, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της τάξης του 0,88 δεν θα μπορέσει να <clears throat> επιτευχθεί. Ταυτόχρονα χώρες ε, που έχουν ανάγκη από βοήθεια ε, συνεχώς αυξάνονται. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το κονδύλι να μην σε και εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης ε, να αναζητηθούν. Παρόμοια ζητάμε να υπάρξει μια συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον έλεγχο η νομική βάση σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται το μέσο για τι μηχανικέ χώρε, θα ε, πέσει στο, θα πέσει στο πλαίσιο της ε, συναπόφαση. Επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταβασική φάση, το δικαίωμα για δημοκρατικό έλεγχο δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω στον κανονισμό, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να δεσμευτεί να δώσει το Κοινοβούλιο τα ίδια δικαιώματα ε, για το τροποποιημένο μέσο και αυτό πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου να εγκρίνει το Κοινοβούλιο επειδή ο κύριος ε, Ντέβα που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα θα μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις σας ε, γραπτός ή στο πλαίσιο διμερών επαφών αν τα μέλη λοιπόν επιθυμούν μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή, αυτό μπορούσε, να επιτευχθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου στην εδρίαση της Επιτροπής μας πριν από την ψήφιση των τροπολογιών. Mr. Berman, you have the floor. Dank u mevrouw de Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι κάτι που μπορούμε να το την συζητήσουμε. Σκοπό έχει να καταπολεμεί τη φτώχεια πρωτίστως και βέβαια μπορούμε να δούμε τι είναι η φτώχεια μετά. Πάντως η Επιτροπή μας πρέπει να δίνει κάποιες εγγύσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προασπίζουμε τον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας και πρέπει να τον διαφεντεύομαι απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή. Ε, ε, παντού τώρα η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια συνδέεται με το ΑΕΠ και όλοι πάνε να πιάσουν το 0,7%. Το 0,7% ε, όμως ε, μειώνεται σε συνάρτηση με το ΑΕΠ που μειώνεται παντού. Τώρα θα πρέπει να αυξηθεί πρέπει να πληρώνουν περισσότερα ε, όλοι για τις πιστώσεις τους, ε, για το εμπόριο κλπ. Πρέπει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να την υπερασπιστούμε τώρα περισσότερο από ποτέ. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την αναπτυξιακή συνεργασία και πρέπει να δαπανώνται τα χρήματα με καλύτερο τρόπο, αλλά όχι να μειωθούν. Δεν πρέπει ο προϋπολογισμός να συρρυκνωθεί, όπως ε, άλλωστε πρότεινε προηγουμένως και ο κύριος Πινκ. Πολλές φορές βλέπουμε πράγματα που μας ξενίζουν. Μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους να φορούν ε, ε, παπούτσια ποδοσφαιρικά ή να είναι ξυπόλυτη. Ε, όλα αυτά είναι δυνατότητες διαφορετικές και πρέπει και εμείς να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι πρέπει να καλύψουμε αυτό το οτιδήποτε υπάρχει στο άρθρο 4. Ευχαριστώ. Πέρα από το θέμα των αναπτυξιακών κονδυλίων από τον DCI, έχουμε την πρόταση αυτή της Κομισιόν για δραστηριότητες που σαφώς δεν καλύπτονται από τους στόχους του DCI. Και είναι σαφές για μένα ότι τα χρήματα δεν μπορεί έτσι εύκολα να τα παίρνουμε και να τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς άλλους από τους αρχικούς. Πέρα από αυτό το θέμα, δεν καταλαβαίνω και πώς μπορεί να γίνεται η ακαθάριση μιας πολιτικής ε, ε, καθών χρόνων έχουμε ας πούμε αναπτυξιακή βοήθεια και υποστήριξη και με τα ίδια λεφτά, λέει η Κομισιόν, ε, πρέπει να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που είναι προς το οικονομικό όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανενός άλλου. Βλέπω πρόβλημα με τη συνέπεια της πολιτικής μας, γιατί εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τα λεφτά από τον DCI που σκοπό έχουν την εξάλληψη της φτώχειας. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτή η συνοχή στην πολιτική που την θέλει η Κομισιόν, πώς θα εξασφαλιστεί. Και άλλες ερωτήσεις. Τι ακριβώς εννοείται με το άλλες δραστηριότητες, μη ODA, τι είναι αυτές, τι δηλαδή δραστηριότητες ε, προβλέπονται πέρα από αυτές που απαριθμούνται. Και επίσης, πώς είναι δυνατόν χρήμα, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δρά προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών εταιριών διαθέτοντας χρήματα που είναι του DCI και μετά δρά προς το συμφέρον συγκεκριμένων εταιριών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πογκάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα πάρω το λόγο για τα νησιά του Ειρηνικού, από τα οποία και προέρχομαι, σχετικά με αυτό το κείμενο που πρέπει να εγκριθεί και να σας πω ότι εκφράζω ιδιαίτερη ικανοποίηση για αυτήν την πρόταση αναθεώρησης που επιτρέπει να αυξήσουμε τους, τις δικιούχες χώρες ε, με την αύξηση του χρηματοπιστωτικού μέσου. Μόνο οι χώρες ΑΚΕ μέχρι τώρα είναι επιλέξιμες για αυτό το μέσο. Οι πανάπτυξη χώρες εκτός ΑΚΕ εντάσσονται μόνο στο σχέδιο για την καταπολέμηση της παινίας. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ως μόνη προτεραιότητα την καταπολέμηση της παινίας. Θέλουν οικονομική και εμπορική ανασυγκρότηση. Θέλουμε λοιπόν και οι αναπτυσσόμενες χώρες να είναι δικαιούχοι του, αυτού του χρηματοπιστωτικού μέσου. Εγώ είμαι Γάλλος Ευρωβουλευτής. Έρχομαι από τις υπερπόντιες γαλλικές περιοχές και θέλω να τονίσω εδώ το καθεστώς ε, της ε, Νέας Καλλιδονίας η οποία την χάνει ειδικού καθεστώτος ως μέλος της Ένωσης. Και στη Νέα Καλλιδονία και στις άλλες υπερπόντιες περιοχές αυτό το οποίο στοχεύεται δεν είναι η καταπολέμηση της ε, παινίας, αλλά η αύξηση του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας. Η αναθεώρηση λοιπόν αυτού του χρηματοπιστωτικού μέσου πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή των υπερποντίων γαλλικών περιοχών στην, στο μέσο αυτό. Η Κομισιόν ζητάει το λόγο. Ο κύριος Μενιέ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αν δεν υπάρχουν άλλα σημεία από τους βουλευτές, εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα σχετικά με τις δημοσιονομικές ε, πτυχές και να απαντήσω αμέσως στον κύριο Πόγκα. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να επεκτείνει το εφαρμοστικό πεδίο που έχουμε από τις, από τις βιομηχανοποιημένες χώρες ε, στις ε, χώρες ε, που εντάσσονται στα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά οι υπερπόντες γαλλικές περιοχές δεν εντάσσονται σε αυτό το μέσο. Τώρα, για τις δημοσιονομικές πτυχές που βρίσκονται και στο επίκεντρο της συζήτησης, αυτής της Επιτροπής, ε, διότι υπάρχει αυτή η αντιμαχόμενη πρόταση της ε, Κομισιόν να επαναχορηγηθούν ορισμένες πιστώσεις, ε, να αναδιερμηθούν μάλλον, με την, διευρύνοντας το εφαρμοστικό πεδίο του μέσου. Όμως θα πρέπει να εξυπακούονται τρεις στόχοι. Οικονομική συνεργασία, την business partnership νομίζω το λένε στα αγγλικά, που θα πρέπει να αποτελούν νομοθετική συνέχεια των δύο προπαρασκευαστικών δράσεων που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο το 2008 και δεν μπορούμε να τραβήξουμε πέρα από το 2009 διότι ισχύουν μόνο τρία χρόνια αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Αφορά κυρίως αναδυόμενες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια συνεργασία πέραν της εκρίζωσης της φτώχειας. Σε δημοσιονομικό τώρα επίπεδο, η Κομισιόν συνεισφέρει για αυτό το κεφάλαιο με 68 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή, την περι... σε αυτή τη διάρκεια. Συνεισφέρει λοιπόν με αυτό το ποσό για να εγγυθεί τη συνέχεια των δράσεων αυτών. Προσθέτοντας και κάτι παραπάνω δηλαδή για να συνεχιστεί το όλο εγχείρημα των τριών ετών. Βέβαια δυστυχώς ήταν μια απόφαση ιδιαίτερα επίπονη για τους επιτρόπους μας και την Κομισιόν. Λόγω δηλαδή της στενότητας της οροφής ε, του πλαφών, δηλαδή του τίτλου 4, δεν μπόρεσε να προτείνει τα 76 εκατομμύρια, όλα μαζί δηλαδή από το περιθώριο του τίτλου 4. Υπάρχει αυτό το impact assessment που συνοδεύει την νομοθετική πρόταση και που αναλύει τις ε, επιλογές. Ε, άλλοι λέγανε 100% από το περιθώριο να χρηματοδοτήσουμε, άλλοι λέγαμε ναι, να γίνει πλήρης αναδιανομή του μέσου για τις βιομηχανοποιημένες χώρες και άλλες λέγανε να έχουμε μία μεικτή κατάσταση με νοπό χρήμα. Εμείς ε, επιλέξαμε αυτή τη λύση διότι έχουμε διάφορες ανταγωνιστικές προτεραιότητες μέσα σε αυτή τη ρουμπλίκα, μέσα σε αυτό το τίτλο 4 και το περιθώριο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Κυρίως άμα δούμε δηλαδή χρηματοδότηση της Παλαιστίνης, χρηματοδότηση των κλιματολογικών αλλαγών κτλ. Η Κομισιόν λοιπόν αποφάσισε να προσεγγίσει το θέμα λέγοντας ότι πρόκειται για μια νέα πολιτική που αποτελεί συνέχεια των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Μια νέα πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναδυόμενες χώρες και να χρησιμοποιήσει αυτό το περιθώριο. Τώρα για τα δύο άλλα κεφάλαια που αφορούν στην παιδεία και τις άλλες δράσεις οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες υπό τον τίτλο «Δημόσια ενίσχυση για την ανάπτυξη. Η Κομισιόν το είχε προβλέψει στην αρχική πρόταση του DCI, αλλά η επιλεξιμότητα περιορίστηκε στα στενά κριτήρια της δημόσιας ε, βοήθειας για την ανάπτυξη. Ε, προβλέψαμε ότι υπάρχει ας πούμε, διασφαλίστη κινητικότητα με προγράμματα όπως το Erasmus Mundus, όπου οι αλλοδαποί φοιτητέ όταν έρχονται στην Ευρώπη είναι επιλέξιμοι για τη δημόσια ενίσχυση για την ανάπτυξη, αλλά τα πανεπιστήμια από όπου προέρχονται δεν είναι επιλέξιμα. Η Κομισιόν θέλησε να το επαληθεύσει, αλλά ο χρηματοδοτικός φάκελος προβλεμόταν σε αυτό το μέσο και θέλει να του προσδώσει σήμερα η Κομισιόν τη, σωστή νομική βάση που έχετε μπροστά σας σήμερα. Τώρα υπάρχει αυτή η φαιά ζώνη Είπαμε τα κριτήρια ήταν βέβαια πολύ καθαρά, αλλά ε, από τεχνικής ε, πλευράς αυτές ε, οι δράσεις, δηλαδή όσον αφορά στην τεχνική υποστήριξη στην Κεντρική Ασία για την ενεργειακή ασφάλεια κλπ. Υπήρχε πρόβλημα, όπως επίσης και σε διάφορες διπλωματικές δράσεις στο Ιράκ και στο Ιράν που δεν είναι επιλέξιμες ως δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη, αλλά εντάσσεται στον DCI. Μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ε, σε δύο-τρεις περιφέρειες. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα ζυγίσουμε. Ήταν μια απόφαση δύσκολη για την Κομισιόν για την ανομή ε, των δημοσίων ενισχύσεων για την ανάπτυξη δεν θέλαμε εμείς να αλλάξουμε ανατολισμό στο χρήμα ε, της αναπτυξιακής βοήθειας ε, για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Αλλά σίγουρευτήκαμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό φάκελο DCI, δεν αλλάζει 17 δις ευρώ Σήμερα ο προγραμματισμός μέχρι το 2013 ξεπερνάει τα 17 δις, πέρα δηλαδή από την αναδιανομή, ξεπερνάμε λοιπόν το κατόφλι αναφοράς και οι επιπτώσεις αυτών των 100 εκατομμυρίων στα τελευταία χρόνια και αν το δούμε στην Κεντρική Ασία και στην Νότια Αμερική είναι, από, ε, είναι 6 εκατομμύρια στην ε, Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Ασία είναι γύρω στα 10-15 το μήνα, είναι 800 εκατομμύρια το χρόνο για την Κεντρική Ασία. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σήμαντες. Τώρα, όσον αφορά στους ε, περιφερειακούς δημοσιονομικούς ε, ε, φακέλους, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα και η Κομισιόν κάθε χρόνο προτείνει στα πλαίσια του προσχεδίου προϋπολογισμού μία χορήγηση πιστώσεων για τον κάθε τίτλο και την τελευταία λέξη την έχει το Κοινοβούλιο. Και πάντα αφήνει η Κομισιόν ένα περιθώριο. Πάντα Λοιπόν, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε κονδύλια, να προσθέσετε ποσά. Ευχαριστώ. Και διατρέχω τον κίνδυνο να είμαι επαναληπτικός. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε με την Κομισιόν. Εμείς είχαμε αυτή τη συζήτηση στην αρχή της χρονιάς. Την ίδια συζήτηση για τη Λατινική Αμερική όταν είπαμε για την ανταλλαγή μεταξύ Αργεντινών και Ισπανών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Αραγώσα. Εμείς ε, χειροκροτάμε ε, που ορισμένα κοινωνικά στρώματα της Βραζιλίας, Αργεντινής, της Χιλής ε, βγαίνουν από το σπέκτρο της φτώχειας. Και λέμε και πανηγυρίζουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας ορίστε τι φοβερή επιτυχία με αυτές οι αναλλαγές. Αλλά είναι σκανδαλώδες εμείς να ζητούμε από τις χώρες εκείνες να πληρώσουν αυτή την ανταλλαγή φοιτητών. Διότι δεν είναι δικιούχοι για αυτές τις ανταλλαγές, αλλά πρέπει από το δικό τους δημοσιονομικό φάκελο να βγάλουμε τα χρήματα για να τα πληρώσουμε. Δεν φτάνουμε καν εμείς οι αναπτυγμένες χώρες αυτό το 0,7% που είχαμε δεσμευτεί να δίνουμε. Και δεν ξέρουμε καν που θα βρεθούν τα λεφτά και με ποιο πρόσχημα θα τα βγάλουμε. Και έστω κι αν είναι 4 με 6 εκατομμύρια το χρόνο, πρόκειται για ένα προηγούμενο και πρέπει να μην δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο. Άσχετα από το αν ο στόχος όπως η ανταλλαγή φοιτητών είναι ένας πολύ ωραίος στόχος και κανένας δεν τον αμφισβητεί. Σταματήστε λοιπόν να ροκανίζετε τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη και βρείτε άλλα κονδύλια να τα φάτε από αλλού υπάρχουν και άλλοι φάκελοι. κυρία Κέλλερ. Η πρόταση αυτή παίρνει ε, αυτές τις παρατυπίες και τους φτιάχνει μια νομική βάση. Ε, πάντως εγώ δεν άκουσα να απαντούνται οι ερωτήσεις μου σχετικά με τη συνοχή με τις άλλες αναπτυξιακές πολιτικές και τι είναι αυτές οι άλλες δραστηριότητες ε,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 Ευχαριστώ Πρόεδρε σε ό,τι φορά την συνοχή. Οι ίδιες υπηρεσίες ε, είναι αυτές που διασφαλίζουν τον προγραμματισμό του μέσου συνεργασίας και αυτή η νέα πτυχή του μέσου. Δηλαδή η συνοχή θα είναι απόλυτη και εδώ πρόκειται για μια περιφερειακή θα λέγαμε, περιθωριακή θα λέγαμε συνεργασία. Μιλάμε για 116 εκατομμύρια τα τέσσερα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο μια συνεργασία τη τάξη του 1,6 δι ετησίω. Το επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας όπου ξεκίνησε το 2007-2008 είχαμε προτείνει να ανοιχτούν κάποια business center στην Ινδία, στην Κίνα και αλλαχού, να υποστηρίξουμε την ψηφιακή τηλεόραση στη Λατινική Αμερική, να προωθήσουμε την ε, ε, διπλωματία στην ε, Ινδία και λοιπά στην Κεντρική Ασία. Εν δεν δεσμεύουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις χώρες ε, προκειμένου να προασπίσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Η συνοχή λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι είναι απόλυτα διασφαλισμένη, είναι οι ίδιες οι μονάδες που εργάζονται υπό την αυτή η γενική διεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να πω προς την Επιτροπή ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να λειτουργούν τα κονδύλια για την ανάπτυξη για τις βιομηχανικές χώρες. Ο προϋπολογισμός είναι ήδη ανεπαρκής για το έργο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το μέσο λοιπόν αυτό είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον, αλλά αυτή η λειτουργία σύμφωνα με το DCI δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτά. Αν δεν επιθυμεί κάποιο άλλο να λάβει το λόγο, επενθυμίζω πως μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες στο κείμενο μέχρι την 15η Οκτωβρίου το μεσημέρι. Και τώρα μπορούμε να εξετάσουμε το τελευταίο σημείο της μεσαίας διατάξεως. Πρόκειται για μια παρουσίαση από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που συστάθηκε το 1951. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. Υπάρχουν πάνω από 50 εθνικές κυβερνήσεις ε, Δήμων, ε, Κοινοτήτων και Περιφερειών ε, που εκπροσωπούνται και αυτό αντιστοιχεί σε 100.000 τοπικές αρχές ε, και αυτοδιοίκησεις που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο αυτό. Σήμερα βρισκόμαστε τον... Ε, έχουμε μάλλον το επικεφαλής ε, των επαφών, των δημόσιων επαφών αυτού του οργανισμού, τον κύριο Φιωρέλη, ο οποίος ε, θα μας ε, κάνει την παρουσίαση της, ε, του δικτυακού τόπου του Συμβουλίου Δημοτικής περιφέρειας της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο έχει χρηματοδοτήσει η Κομισιόν και έχει ως στόχο την αναζήτηση εταίρων για την εξέταση μιας σειράς προβλημάτων. Κύριε Φιωρέλη, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή στο θέση θα ενδιαφέρει πάρα πολλά άτομα που εργάζονται μέρη συνεργασία. Δέκα λεπτά μου δώσατε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έφτασα λίγο νωρίτερα γιατί μπορούσα να παρακολουθήσω τις ε, συζήτησε. Τις Όταν μιλήσατε για τα μη κρατικά προγράμματα, άκουσα να μιλάμε για μη κυβερνικέ οργανώσεις, αλλά δεν άκουσα να αναφέρεστε καθόλου σε δήμους ε, και κοινότητες. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Concord, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστώ για μια δεύτερη φορά που μας ε, επιτρέπεται να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, διότι το μήνυμα θα ήθελα να περάσει. Είπατε λοιπόν ότι εμεί δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή οργάνωση, είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Δημιουργήσαμε αυτό το δικτυακό τόπο για τι πόλει του Βόρεια και του Νότου, ε, διότι εμεί ε, δημιουργήσαμε και την έννοια της ε, αδελφοποίησης στην Ευρώπη το 1951 ε, βλέπετε εδώ στην, την αριστερή πύλη και δουλεύουμε με πάνω σε αυτό. Το γραφείο του Λουί Μισελ ήρθε να μας συναντήσει και μας είπε ότι μια που δουλεύετε κάτι τέτοιο θα μπορούσατε να κάνετε κάτι παρόμοιο για την ανάπτυξη, ανάπτυξη βορανότου αποκεντρωμένη μόνο και μόνο, και μόνο για τις πόλεις. Και εμείς απάντησαμε ναι, διότι θα ήταν πιο εύκολο παράδειγμα ε, δεκτή όπως ε, από το τίποτα, να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Ελπίζω να λειτουργήσει η σύνδεση. Φτιάξαμε λοιπόν ένα τόπο 25, σε 25 γλώσσες με αυτόματη μετάφραση και για το τμήμα Βορανό το να είναι τετράγλωσσος διότι δεν είχαμε πολλά χρήματα, είχαμε μόλις 20.000 ευρώ στη διαθεσή μας και είπαμε ότι με τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα πορτογαλικά καλύπταμε σχεδόν όλη την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Δεν θα μακρηγορήσω. Περί τίνος ακριβώ πρόκειται. Υπάρχουν δύο τμήματα, ένα που είναι ιδιαίτερα παιδαγωγικό και αφορά τις ε, την τοπική αυτοδιοίκηση, εξηγώντα του ε, τι σημαίνει η αποκεντρωμένη συνεργασία, ποιο ε, λαμβάνει μέρο, σε ποιον μπορώ να αποτανθώ, είναι αυτό το παιδαγωγικό που θα λέγαμε. Και ένα ενδιαφέρον κομμάτι για τους Δήμους και τις τοπικέ περιφέρειες, ε, θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος γραφείου συνοικεσίων για, τις, ε, για τους Δήμους και τις περιφέρειες και κοινότητες. Ε, οποιαδήποτε πόλη λοιπόν, βορρά του νότου, μπορεί να συμπληρώσει ένα έντυπο και να αφήσει ένα, μια, μια αναγγελία πάρουμε τον πολυμαραντή του στην Νιγερία ότι με κάποιες πληροφορίες, με έναν χάρτη που μας επιτρέπει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η πόλη και ότι αναζητάει εταίρους ε, για μια αποκεντρωμένη συνεργασία κλπ. Είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην πόλη αυτή διότι αναζητούν ε, πολλούς εταίρους. Τους ζητάμε επίσης ε, τι μέγεθος πόλη ψάχνεται διότι μια πόλη 100.000 κατοίκων διαφέρει τι από μια πόλη 5 εκατομμυρίων και τι ενδιαφέρεστε για την οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντικά θέματα, διαχείριση αποβλήτων. Τη λοιπόν που αυτή η πόλη Μαραντή έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, δεν βγαίνει κατευθείαν online, εμεί θα ελέγξουμε αν πρόκειται για μια αληθή ή όχι ε, αναζήτηση και ταυτόχρονα όταν μπει στο σύστημα Μεταφράζεται σε τέσσερις γλώσσες. Θα μπορούσα να σας μιλάω για τουλάχιστον μια ώρα, εμπεστώς έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, πάντως καταλάβατε το, το θέμα. Σας πω για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Αυτό εντάξει είναι μια ιστοσελίδα που μπορεί να ελέγξετε. Αυτό η ε, ιστοσελίδα ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και παρατηρούμε ότι σας έχουμε ανάγκη. Πρέπει να γνωρίσουν ε, οι περισσότεροι βουλευτές το τι συμβαίνει. Ε, οι ευρωβουλευτές περισσότεροι ξεκίνησαν από την τοπική αυτοδιοίκηση, δούλεψαν σε επίπεδο πόλεων, δήμων και κοινοτήτων. Θα δούμε σε κάποιους οι οποίοι έχουν κάποιες ε, γνώσεις πάνω στο θέμα, έχουν κάποιες χορδές που μπορούμε να θίξουμε Νομίζω λοιπόν πως ε, αξίζει τον κόπο για μας, εμείς είμαστε ένας μη κυροσκοπικός οργανισμός, αλλά για τις πόλεις του ώρα και του Νότου, γεγονός ότι ε, γνωστοποιούν πως υπάρχει ένα, μια, ένας διεκτυακός τόπος μέσω του οποίου μπορούν να στενηθούν πόλεις ε, και να δημιουργήσουν εταιρικέ σχέσεις, επαφές και αδελφοποίησης αξίζει τον κόπο. Εμείς στον οργανισμό έχουμε δραστηριοποιηθεί εδώ και χρόνια. 60 χρόνια ε, ε, ε, είναι από τότε που έχουμε συσταθεί. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια πλατφόρμα για τις τοπικές αρχές, για τη συνεργασία. Αυτό είναι ένα από τα μέσα που έχουμε διάθεσή μας. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να βασιστούμε στην υποστήριξή σας προκειμένου να γίνουμε γνωστοί τόσο στο βαρός και στο νότο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων. Ευχαριστώ, δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Εάν euh, δεν επιθυμεί κάποιος να λέει το λόγο, α, παρακαλώ. Λίγα λόγια μόνο. Εγώ έρχομαι από μια χώρα απόλυτα αποκεντρωμένη όπως η Ισπανία. Και πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω με μία ε, θετική εμπειρία για τη συνεργασία, για την αναπτυξιακή συνεργασία μέσα από ενδιάμεσες, ε, ε, ενδιάμεσους θεσμούς που δεν είναι η κεντρική κυβέρνηση. Στην Ισπανία μιλάμε για αυτόνομες κοινότητες, είναι τα λέντερ, τα κρατήδια στη Γερμανία περιφέρειες ονομάζονται αλλού. Τέλος πάντων, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές αρχές. Είναι μια εμπειρία πολύ θετική, διότι μόλις, όπως ανέφερε τώρα ο εμπειρογνώμονας, γίνεται άμεση συνεργασία μεταξύ οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δημαρχείου με δημαρχείο. Μπορούν να, γίνουν, να ανταλλάσσουν θετικές πρακτικές, ε, πειράματα που δούλεψαν και μπορούν να υποφεληθούν ε, ε, όλοι. Έτσι λοιπόν, υπησέρχεται και ο παράγοντας εξειδίκευσης σε συγκεκριμένες περιοχές, σε δήμους, σε κοινότητες από χώρα σε χώρα. Δηλαδή υπάρχει μία διαβάθμιση από την κρατική συνεργασία στη συνεργασία σε άλλα επίπεδα. Εκείνο που πρέπει να εγγυθούμε είναι να μην υπάρχουν επικαλύψεις των ιδίων δράσεων, δηλαδή σε κρατικό επίπεδο, σε ενδιάμεσο ή σε τοπικό επίπεδο. Αν αποφύγουμε όμως αυτό το πρόβλημα, αυτό το οποίο κατακτάμε από την αποκέντρωση της αναπτυξιακής βοήθειας είναι απόλυτα θετικό. Euh, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire euh, Moins d'une minute, Madame la Présidente. Euh, Merci. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Εγώ συνεργάζομαι με μία ένωση που λέγεται Mondial de Ville, όπου ακριβώς γίνεται η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά τώρα για την αποφυγή της επικάλυψης εννοείται. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως, διότι πρόκειται για μεμονωμένες δράσεις μίας πόλης που ψάχνει έναν άλλο εταίρο από την άλλη μεριά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι μια πολύ καλή Μια πολύ καλή πρωτοβουλία όταν ένας δήμαρχος επιλέγει να συνεργάζεται με μία και μόνη πόλη. Πάντως ε, σας λέω ότι σε αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος επικαλύψεων. Κυρία Βέρνμαν Κρόου, θέλετε το λόγο. Από τα τέλη του 2008 η Κομισιόν δεσμεύτηκε σε μία αναγνώριση του ρόλου ε, της ε, περιφερειακής ε, και των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην συνεργασία και στην ανάπτυξη. Αναγνωρίστηκε δηλαδή ο ρόλος των τοπικών αρχών με τη συνεισφορά τους δηλαδή ως χρηματοδότες Άρα και στη συνεισφορά τους ε, σε, στο θέμα της ε, διαχείρισης του ύδατος, της ε, υγειονομικής παρέμβασης, της ε, διακυβέρνησης κλπ. Και εμείς δεν θέλουμε μία καταναγκαστική συνεργασία της τοπικής αυτοδίκησης, αλλά θέλουμε να έχουμε διάφορα μέσα, προτείνουμε διάφορα εργαλεία για να υπάρχει μία ορθολογικοποίηση αυτής της συνεργασίας και διερευνούμε εμεί τρει ε, υποθέσεις. Πρώτον, η υλοποίηση ενός Άτλαντα για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Γιατί πρέπει να το λάβαμε υπόψη μα αυτό όταν φτιάχναμε την ανακοίνωσή μας όπου δεν είχαμε μία πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, στην Ευρώπη πρόκειται πάνω από 80.000 ε, ε, μονάδες δύσκολο είναι λοιπόν να ξέρει κανείς τι κάνουν οι μεν και οι δε χρειάζεται λοιπόν ένας άτλαντας σχετικά με τις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συνεργασία και την ανάπτυξη τον ε, συντάσσουμε σε αυτή τη φάση τον Άτλαντα και ελπίζουμε να τον έχουμε και στη διάθεσή μας μέχρι τα τέλη της χρονιάς το Δεκέμβριο. Δεύτερη υπόθεση προβληματισμού είναι ο, διαπιστώσαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δραστήρια στην αναπτυξιακή βοήθεια και σε μία φάση όπου η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας βρίσκεται στην καρδιά ε, της κάθε συζήτησης θελήσαμε να, ε, να ισχυροποιήσουμε τον διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό οργανώσαμε και τη συνέλευση της ΑΣΥΣ εδώ στις Βρυξέλλες ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και θελήσαμε να έχουμε την αποκεντρωμένη συνεργασία με πρωτοβουλίες που όπως τις παρουσίασε και το ΣΕΣΕΡ σήμερα με την ιδέα με την ιδέα που στον καιρό της ονομαζόταν αδελφοποίηση μεταξύ των διαφόρων πόλεων. Ε, θέλουμε λοιπόν να έχουμε συνεργασία μεταξύ των πόλεων και με τη βοήθεια της Επιτροπής των Περιφερειών θέλουμε να ξεκινήσουμε έναν πραγματικό διάλογο και να ανασύρουμε όλα τα πλεονεκτήματα της συνεισφοράς, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Περιφερειών, με το ΣΣΕΡΕ και όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης